Bueno, si les parece, comenzamos. Luego se quejan del presidente. Λοιπόν, αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε, γιατί μετά παραπονιέστε για τον πρόεδρο. Με 20 λεπτά καθυστέρηση ξεκινάμε. Ο κ. Στίβενσον έχει το πρώτο θέμα σήμερα σε διάδοξη. Πολύ ωραία. Bueno, pues si les parece, como no está el señor Stevenson y la señora Rod... Λοιπόν, ο κ. Στεφανσόν δεν είναι εδώ, κύριε είναι. Συμφωνείτε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη για να μην χάνουμε χρόνο και να περάσουμε στο σημείο 11. Και κατόπιν δούμε το 10 για να μην χάνουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, ποιο θέλει να μιλήσει, να μου πείτε από τώρα και να περιοριστούμε στο δυνατό περισσότερο γιατί πραγματικά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Comenzamos con Con el punto número 11, eh, ya hemos intercambiado punto de... Λοιπόν, ας περάσουμε στο σημείο 11. Και τώρα κατευθείαν να δώσω το λόγο στην κυρία Ρόντουστ για να μας μιλήσει για το θέμα της ε, στο πλαίσιο της Μεσογείου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συμφωνώ να αλλάξουμε την σειρά των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Βρίσκω ωστόσο κρίμα που είναι τόσο λίγες και τόσο λίγοι παρόντες. Σε ποιον θα τα πω δηλαδή εγώ. Ελπίζω οι συνεργάτες των βουλευτών να τους τα μεταφέρουν. Συμφώνησα με τους και οδησίγητες να μιλήσουμε σήμερα ειδικά για την Μεσόγειο και τις επιπτώσεις της μεταρρυθμίσεως. Η Μεσόγειος που είναι και το προβληματικό πεδίο ας πω έτσι, της κοινής ελευτικής πολιτικής είναι η άγρια δύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έλεγχος στην Αλία και ως λόγο αναφέρουν πολλοί τον, την ύπαρξη πολλών, μη, ε, πολλών χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα ψάρια ωστόσο ψαρεύονται μέσα στην αποκλειστική ζώνη των 12 μιλίων, άρα δεν τα μοιράζονται αυτά με χώρες όπως η Λιβύη, την Ισία κλπ. Εν πάση περιπτώσει από το 2006 γίνεται μια προσπάθεια να επιτευχθεί κάτι. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις το Συμβούλιο ενέκρινε και ψήφισε τον κανονισμό για τη Μεσόγειο, που δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος. Παρ' όλα αυτά οι χώρες μέλη καλούνται να, και υποχρούνται να κάνουν προγραμματισμό αλλά έχουν μεγάλη δυσκολία με την τήρηση των σχεδίων αυτών. Η εφαρμογή της κοινής αλληλευτικής πολιτικής δεν είναι καθόλου καλή. Δεν υποβάλλουν σχέδια διαχείρισης οι χώρες μέλη. Όλες οι χώρες μέλη θίγονται. Ορισμένες ε, δεν... Ε, αυτό αφορά μάλλον όλες τις χώρες μέλη. Ορισμένες δεν κάνουν τίποτε, άλλες κάνουν ανεπαρκή πράγματα. Από τη σκοπιά μου ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πρώτον να ασκήσουμε πίεση ώστε να εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμός. Ίσως χρειαστεί να ε, εγκρίνουμε κάποια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία ή ένα ψήφισμα. Αυτό βέβαια είναι ευθύνη κυρίως του Συμβουλίου. Εφόσον όμως το Συμβούλιο Υπουργών ούτε καν τις δικές του αποφάσεις δεν εφαρμόζει, ε, βεβαίως θα διαφορήσει πλήρως για τις δικές μας αποφάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεύτερο, να διατυπώσουμε τις δικές μας ιδέες. Πώς θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνει η διαχείριση της αλίας στην Μεσόγειο. ώστε να βελτιωθεί ο κανονισμός. Η κοινή αλληλευτική πολιτική και η μεταρρύθμισή της θα πρέπει να δώσει τις σωστές βάσεις. Ποια πράγματα πρέπει να λάβουμε υπόψη στον κανονισμό θα πρέπει να δώσει προσανατολισμούς για το πώς θα πρέπει να είναι ο κανονισμός για την Μεσόγειο. Ο βασικός κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα εμπόδια. Η κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεκτική. Χρειαζόμαστε ένα κοινό πλαίσιο το οποίο να περιλάβει και την Μεσόγειο. Ταυτόχρονα το πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Τα προβλήματα στην εφαρμογή στην Μεσόγειο δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν σε πολύ περιορισμένες φιλοδοξίες στη μεταρρύθμιση μας. Όλα αυτά είναι μια σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο με λόγια. Πρέπει να εργαστούμε καθαρά, ξεκάθαρα δηλαδή, και ορισμένοι φοβούνται ότι ο νέος κανονισμός θα υπερεπιβαρύνει την ε, αλληλεία στη Μεσόγειο. Αυτό είναι κατανοητό. Αν όμως η Μεσόγειος θέλει να προχωρήσει σε μια βιώσιμη αλληλεία, θα χρειαστεί να κάνει περισσότερα βήματα. Και διότι η Μεσόγειος υφίσταται τέτοια καταστροφική υπεραλίευση και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Στις άλλες θάλασσες υπάρχουν κάποια μέσα για αντιμετώπιση της υπεραλίευσης. Πού βρίσκονται τώρα συγκεκριμένες δυσκολίες. Ο κανονισμός για το MSI δίνει σωστούς κανόνες για τον Ατλαντικό και για τη Βαλτική είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ότι αυτά πρέπει να γίνουν δηλαδή με προσαρμογή των ποσοστώσεων. Για την Μεσογείο δεν υπάρχουν ποσοστώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την υπερβάλλουσα αλληλευτική ικανότητα. Και εδώ έχουμε ένα μέσον, τα TFC δηλαδή, για την μείωση της περιβάλλουσας αλληλευτικής ικανότητας. Όπου υπάρχουν ποσοστώσεις, το εργαλείο αυτό λειτουργεί. Εδώ όμως δεν λειτουργεί, διότι δεν υπάρχουν ποσοστώσεις για να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι λάθος, διότι βασικός στόχος του κανονισμού θα πρέπει να είναι να βάλει βασικούς στόχους με προθεσμίες και να χορηγήσει τα κατάλληλα μέσα. Η εφαρμογή θα γίνει επιτόπου, καθώς και η περιφερειοποίηση. Έχουμε υποβάλει κάποιους στόχους για τη Μεσόγειο, αλλά δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα, τα, εργαλεία. Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί μας από τη Μεσόγειο θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, θέλουν να αντιδράσουν στην υπεραλίευση και ότι είναι διατεθειμένοι να πράξουν περισσότερα από ό,τι πράττουν οι κυβερνήσεις τους. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε την ιδιαίτερη αυτή κατάσταση της Μεσογείου. Αφενός, για το μεγάλο γενικό πλαίσιο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μέσα στον βασικό κανονισμό, είναι να προσαρμόσουμε τις προθεσμίες. Σε όλες τις περιφέρειες όπου η κατάσταση είναι περιπλοκότερη, όπου χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία λύσεων, θα πρέπει να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο. Περισσότερο χρόνο για την ε, εφαρμογή, για παράδειγμα, της απαγόρευσης, της απόρριψης στην θάλασσα των ανεπιθύμητων ειδών. Επίσης για τα TFC και καθώς επίσης και για την πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα. Θα πρέπει να βάλουμε και άλλους στόχους, για παράδειγμα για την μέγιστη βιώσιμη απάδοση. Πρέπει να δούμε πόσα ψάρια μπορούν να ψαρεύονται μακροπρόθεσμα, μπορούμε να βάλουμε και ανώτατα επιτρεπόμενα αλλιεύματα για την ε, ε, Μεσόγειο. Άλλη δυνατότητα θα ήταν να δημιουργήσουμε ζώνες που να είναι ελεύθερες από ε, αλία. Να μην επιτρέπεται δηλαδή απολύτω καμία αλία. Για παράδειγμα στου τόπους όπου αναπαράγονται τα ψάρια. Εκεί μετά για τα υπόλοιπα μπορούν να βγουν και τα πρώτα τάκ. Όλα τα μέτρα που περιλαμβάνουν και ξεκάθαρες προθεσμίες μέσα στον κανονισμό δίνουν κάποια δυναμική στις αλλαγές αυτές εάν πρόκειται το 2018 να θεσπιστεί ένα ανώτατο επιτρεπόμενο αλίευμα, θα έχουν και περισσότερα κίνητρα οι χώρες μέλη, ώστε μέχρι τότε να λάβουν κάποια μέτρα. Χρειαζόμαστε τέτοιους μακροπρόθεσμους στόχους για να έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του κανονισμού για τη Μεσόγειο πριν από τις προθεσμίες αυτές. Αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο μεγάλο έργο μας μετά από την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και να βάλουμε μέσα και να εφαρμόσουμε τη νέα μας αρχή της περιφερειοποίησης. Εγώ είμαι βόρεια, δεν είμαι ειδική για θέματα της Μεσογείου. Έχω όμως πολλούς συναδέλφους από, την, ε, από χώρες της Μεσογείου στην πολιτική μου ομάδα που έχουν συνεργαστεί στενά μαζί μου και εξακολουθούν να συνεργάζονται. Θα εκπονήσουμε λοιπόν νομίζω ορθή πρόταση για τη Μεσόγειο. Και ευχαρίστω να ακούσουμε και από εσά, του υπολείπου συναδέλφου δηλαδή από άλλε πολιτικέ ομάδε, τι προτάσει σα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και βεβαίως μακρηγόρησα κάπως, αλλά ήταν σημαντικό το θέμα. Η κυρία Λόβιν. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο πραγματικά να κάνουμε την ξεχωριστή αυτή συζήτηση για τη Μεσόγειο. Παρόλο που και εγώ εκφράσω τη λύπη μου που είναι τόσο λίγα μέλη παρόντα. Και μάλιστα από μεσογειακέ χώρε δεν είναι κανένα, μόνο ο κύριο Μιλάνα. Ναι, ναι, σας είδα και είπα το όνομά σας. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό του θέματος. Η κυρία Ροντούστ μίλησε για το τραγικό γεγονός ότι ο κανονισμός για τη Μεσόγειο δεν έχει καν εφαρμοστεί. Οι χώρες μέλη δεν υποβάλλουν τα σχέδια διαχείρισης και πολύ λίγα κινούνται, πολύ λίγα πράγματα κινούνται στην Μεσόγειο. Υπάρχει ένας δισταγμός από ορισμένες από τις χώρες μέλη της Μεσογείου. Δεν αρνούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν τα σχέδια διαχείρισης τα οποία αποτελούν μέρος της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Έχουμε και μια τρομερή έλλειψη δεδομένων από την περιοχή της Μεσογείου και σε ό,τι αφορά τα αποθέματα και σε ό,τι αφορά τα είδη, καθώς και την αλλιευτική προσπάθεια και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να τεθεί ως θέμα αφού οι χώρες που θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο για μέτρα στήριξης από το IMF e είναι ορισμένες από τις χώρες αυτές. Αν λοιπόν κανείς δεν σέβεται τους κανόνες της κοινή ελευτικής πολιτικής, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλι... Ε, Θάλασσας και Αλίας. Αυτό είναι το αντικίνητρο που πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο δικαιώματα και υποχρώσεις. Έτσι λοιπόν, ανεπάρκεια δεδομένων είναι από τα πιο σημαντικά εμπόδια για την διαχείριση ιουδήποτε είδου ψαριού στη Μεσόγειο και είναι κάτι το οποίο οφείλει να αντιμετωπιστεί με τρόπο σαφή και εξειδικευμένο. Η διαχείριση των αποθεμάτων, εφόσον δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται, πώς θα γίνει στη βάση της μέγιστης ε, βιώσιμης απόδοσης. Άρα αυτό είναι το νούμερο ένα. Πρέπει να έχουμε πλήρη δεδομένα. Μιλούμε για περιφερειοποίηση. Το περιφερειακό συμβουλευτικό όργανο είναι πολύ χαμηλο προφίλ ακόμα. Η ιδέα περιφερειοποίησης από την πλευρά της Κομισιόν είναι ότι οι ίδιες οι περιφέρειες θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, θα καταθέσουν προτάσεις. Εγώ αναμένω και το ΡΑΚ, να, το Μεσουριακό ΡΑΚ δηλαδή, να δραστηριοποιηθεί. Για, παράδειγμα της Βαλτικής ανέλαβε πρωτοβουλία να προσκαλέσει τις χώρες που βρέχονται από τη Βαλτική να προσέλθουν σε ε, τράπεζα, σε διαπραγματεύσεων να συζητήσουν πώς βλέπουν τη συνεργασία αυτή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για την Μεσόγειο. Είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα κάνει όλα συγκεντρωτικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την περιφερειοποίηση. Διότι είναι και διαφορετικές οι γεωγραφικές και άλλες συνθήκες για τις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες. Είναι σημαντικό για όλες τις θάλασσες να φτιάξουμε ειδικέ προστατευμένε ζώνε σε όλε τι ευρωπαϊκέ θάλασσε, όπου να μην επιτρέπεται η αλία. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία, στον κύριο Μιλάνα, ήρθαν ορισμένοι βουλευτέ με κάποια καθυστέρηση. Κάποιο είπε έξω ότι ξαναρχίζει η συνεδρίαση στι 10.30. Ε, Αυτό ήταν βέβαια λάθος. Ίσως αυτό εξηγεί για ποιο λόγο ήρθαν με κάποια καθυστέρηση ορισμένοι βουλευτές. Εάν το ήξερα αυτό θα περίμενα βέβαια μέχρι και μισή, αλλά κανένας δεν μου είπε ό,τι είχε πει στους ε, βουλευτές ότι θα αρχίζαμε πάλι στις 10.30. Και εξηγώ ότι επειδή ο κύριος Στίβενσον δεν ήταν παρόν, πιστεύω ότι θα αρχίζουμε και μισή, αρχίσαμε με το 11 αντί με το 10 επειδή ήταν παρούσα η κυρία Ρόντου. Ε, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, υπήρξε κάποια παρανόηση και αυτό είναι ο λόγος που ε, συνέβη αυτό. Κύριε Μιλάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πλαίσιο που προτείνει η κυρία Ρόντουστ, όπως εξήγησε και η Ισαβέλα, είναι το πλαίσιο της Μεσογείου. Η εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο ε, είναι κάτι που παρατηρείται. Πρέπει να σκεφτούμε ότι εγκρίθηκε χωρίς τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου με ε, συμφωνία μεταξύ των κρατών ε, και μάλλον κυριάρχησαν λογικές ε, που δεν ε, σεβάστηκαν την κατάσταση στη Μεσόγειο. Υπάρχουν κάποιες ε, διαφοροποιήσεις και ποικιλομορφία, αλλά φυσικά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τη μη εφαρμογή. Ο κανονισμός για τον έλεγχο στην Ιταλία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ακριβώς γιατί έχουμε 800 σημεία από όπου ε, όπου έχουμε αποβίβαση και ε, εκφόρτωση. Και μπορεί να έχουμε εκφόρτωση λίγων ε, κιλών από ένα σκάφο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτές τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη Μεσόγειο και να λάβουμε υπόψη αυτές ε, τις ιδιαιτερότητες ε, και έχουμε μία αλία πολλών ειδών και προσπαθούμε μόνο να την ελέγξουμε με τον έλεγχο των ε, αλευτικών εργαλείων. Όμως κάτι τέτοιο μπορεί να δώσει μεγάλο χώρο στην παράνομη αλία. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε σε μία προοπτική και να επιτρέψουμε στη θάλασσα να εξακολουθεί να αποτελεί πόρο. Νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση που προτείνεται. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτό το κανονισμό και ίσως θα έπρεπε να οικοδομήσουμε κάποιες συνθήκες ε, έτσι ώστε ε, στη μεταρρύθμιση σήμερα να μπορεί να προβλέπονται οι συνθήκες που πρέπει να επαληθεύονται. Τώρα, ε, για την περίοδο αξιολόγηση ήταν ετη δηλαδή αν είχε τη θέση ισχύ το 2010, το 2013 θα πρέπει να γίνει ο έλεγχο. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο από την πλευρά της Επιτροπής να σκεφτεί, να ε, εξετάσει κάτι τέτοιο, όχι το 2013, αλλά ένα χρόνο πριν. Και να πω κάτι άλλο που πιθανότατα επισέρχεται εδώ στον προβληματισμό στη Μεσόγειο. Έχουμε κοινού κανόνε, αλλά δεν είναι όλοι η Μεσόγειο ίδια, δηλαδή υπάρχουν τρομερέ διαφορέ. Αυξήνο πόντο. Ο αυξήνο πόντο έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση και διαθροτική και για το είδο τη αλία και διαφέρει εντελώς από την υπόλοιπη Μεσόγειο. Η Αδριατική στην Αδριατική το ίδιο ισχύει. Διαφέρει πάρα πολύ η θάλασσα αυτή από τις υπόλοιπε και δεν μπορούμε εκεί να εφαρμόσουμε τα ίδια χαρακτηριστικά για τα λευτικά εργαλεία σε μια θάλασσα που έχει 800 χιλιόμετρα μόνο παραλίας και μεσαίο βάθος και φτάνουμε στα 10 μέτρα βάθος σε ένα χιλιόμετρο από την όχθη και από την άλλη πλευρά έχουμε ε, ε, κάθετα βάθη ε, στο Τρινικό Πέλαγος. Έτσι λοιπόν έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη μία θάλασσα στην άλλη. Το λέω αυτό γιατί πράγματι θα πρέπει υπεύθυνα να θέλουμε να γίνει βιώσιμη ελεία στη Μεσόγειο να... Ε, αν δεν θέλουμε πλέον να αλλιεύονται υπερβολικά το 80% των αποθεμάτων, βέβαια υπάρχουν οι έλλειψη στοιχείων για την επαλήθευση αυτού. Ας προσπαθήσουμε όμως να ε, βρούμε τις ιδιαιτερότητες στη Μεσόγειο. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Εγώ νομίζω ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, αλλά εμείς θα πρέπει όχι ίσως να σκεφτούμε ένα και μόνο κανονισμό, αλλά να έχουμε διαφορετικές στρατηγικές, μία, για τη στρατηγική, μία στρατηγική για τον Ευξηνοπόντο, μία για την Αδριατική και άλλη στρατηγική για την υπόλοιπη Μεσόγειο, παραδείγματο χάρη. Η Αδριατική είναι πιο μεγάλη από τη Βαλτική, να το έχουμε αυτά κατά νου. Δηλαδή υπάρχουν και στενά στη Μεσόγειο, αλλά υπάρχουν και τεράστιοι ανοιχτοί χώροι στη θάλασσα. Αυτό το συζητήσαμε μακρόν ε, και με την εισηγήτρια όταν ε, εκπονούμε το κείμενο, όταν εκπονήσουμε το κείμενο πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ιδίω για τη Μεσόγειο πρέπει να εισαγάγουμε καινοτόμους μηχανισμούς. Ιδιαίτερα καινοτόμους και θα αναφέρω ένα. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένας ε, περιορισμός, ένα όριο στην ε, μεταρρύθμιση, είναι ότι ασχολούμαστε με τους ελείς, με τα σκάφη, με τα ίδια ελίας, αλλά δεν ασχολούμαστε καθόλου με τη θάλασσα. Δηλαδή, ο περιέκτης δεν είναι αντικείμενο πολιτικών επιλογών στη μεταρρύθμιση θάλασσα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη θάλασσα, πιστεύω, ότι ιδίω στη Μεσόγειο, εμείς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο να περιορίζουμε τα όσα παίρνουμε και αυτό φυσικά πρέπει να το κάνουμε, αλλά πρέπει να οικοδομήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να παράγει περισσότερο η θάλασσα με δράσεις που να συνοδεύουν και ένα τρόπο οργάνωσης ε, της οδειάς, δηλαδή να έχουμε και πολύ αυστηρούς ελέγχους, αλλά να οδηγήσουμε τη θάλασσα στο να παράγει περισσότερα. Ποια είναι μια πολύ απλή ιδέα, να υλοποιήσουμε ένα πραγματικό δίκτυο non-fishing area, δηλαδή ε, για περιοχές όπου για μία περίοδο ενός μήνα ή για δύο μήνες, όχι μόνο όμως για τις μικρές περιόδους, αλλά για μεγαλύτερες, να, ε, να έχουμε, παραδείγματος χάρη, περιόδους απαγόρευσης μέχρι και τρία έτη, έτσι λέει, ώστε να βοηθάμε τη θάλασσα να παράγει περισσότερο. Αυτό το όραμα δεν αφορά βέβαια μόνο τη Μεσόγειο, αλλά αφορά και την ε, συνολική μεταρρύθμιση της κοινής ελευτικής πολιτικής, αλλά γιατί η Μεσόγειο είναι επιτακτική ανάγκη ε, τα πειράματα που έγιναν σε ορισμένες Ιταλικές περιοχές μας απέδειξαν ε, ότι είναι πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή, αν έχουμε απαγόρευση αλίας ε, σε κάποια χρόνια, είδαμε ότι η θάλασσα αποκρίθηκε και παρήγαγε πολύ περισσότερο. Πρόκειται για μία μέθοδο εναλλακτική στο MSY, γιατί έχουμε μία οικοσυστημική προσέγγιση στο ζήτημα δεν συνδέεται αποκλειστικά με την αξιολόγηση, με αυτό που μπορούμε να αλλιεύσουμε, αλλά ουσιαστικά συνδέεται με δράσεις πολιτικές και προγραμματικές που επιτρέπουν στη θάλασσα να παράγει περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη Μεσόγειο και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε και για τις υπόλοιπες ακτές μας. Και τελευταίο θέμα αφορά την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Εγώ πιστεύω πως αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει μόνο μία μικρή τροποποίηση ή μία μικρή πρόταση στο βασικό κανονισμό. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, και κλείνω πρόεδρε, οι συντονιστές να αντιμετωπίσουν το θέμα με έναν ειδικό τρόπο, δηλαδή ε, σε ένα ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τη Μεσόγειο που να μπορούσε να προβλέψει αυτά τα τρία πράγματα που εγώ μόλις πρότεινα και θα συνοψίσω για να είμαι ακριβής. Καταρχήν, να έχουμε πρόβλεψη των εξολογήσεων για τις επιπτώσεις του κανονισμού για την δηλαδή να, μάλλον, να το κάνουμε νωρίτερα, το 12 για το 13, συγκεκριμένη στρατηγική για την Αδριατική και για τον Αυξηνό Πόντο, με δύο κοινοβουλευτικέ πρωτοβουλίε να προτείνουμε στην Επιτροπή μια συγκεκριμένη οδό που πρέπει να διατρέξει και γιατί όχι μια ε, ρυθμιστική αναθεώρηση. Αν εμεί δεν το κάνουμε αυτό, ενώ θα υλοποιούμε τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΛΠ, ε, πιθανότατα ε, θα έχουμε ε, ανατρέψει την προοπτική για τη θάλασσα αυτή, αν το κάνουμε αυτό. Και τέλος πρέπει να συσταθεί μια στρατηγική από την ε, πλευρά της Επιτροπής ε, έναντι των χωρών της Βόρειας Αφρικής. Και εν μέρει από ό,τι απομένει από τα πρώην Βαλκάνια, αλλά και έναντι και της Τουρκίας και της Ρωσίας γιατί αυτή η θάλασσα έχει μια τέτοια συνέχεια και αν δεν υπάρξει συντονισμός, ε, οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε εμείς για τη διάσωση θα πάει εις μάτιν. Ε, γιατί ξέρετε είμαστε πάρα πολύ κοντά από τη μια στην άλλη και ε, δεν θα υλοποιηθούν οι προσπάθειές μας αν δεν δράσουμε όλοι μαζί. Κυρία Πατράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το σημερινό μας ε, θέμα θα αρχίσω λέγοντας ότι ανέκαθεν υποστήριζε την, την περιφερειοποίηση. Γι' αυτό τον λόγο η κατάρτιση ειδικών σχεδίων ε, για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι ο σωστός δρόμος κατά τη γνώμη μου για να προχωρήσουμε. Δεν ε, έχω καμία αντίρρηση σε σχέση με αυτά που είπαμε για τη Μεσόγειο. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και ευθύνομαι στην κυρία Ρόντουστ. Δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Αναφερθήκατε στο αν ε, μπορούμε ή πρέπει να ε, ε, προσδιορίσουμε συγκεκριμένες ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, δηλαδή για τους αλληλείς της περιοχής εκείνης και μόνο. Μόνο δηλαδή οι αλείς αυτών των περιοχών θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις συγκεκριμένες ε, αλλιευτικές ζώνες. Αυτό εννοούσατε και ε, αν ναι ε, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες και θα ήθελα να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα ποια θα είναι τα κριτήρια για την επιλογή και τον προσδιορισμό, την οριοθέτηση μάλλον αυτών των περιοχών. και γενικότερα σε σχέση με τα αλλιεύματα και τις εξόχους κεντρές ε, περιοχές ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αριοθετούνται οι ευαίσθητες από βιολογική σε πλευρά σε περιοχές ε, διότι ανεξαρτήτως των μιλίων και της απόστασης από την ακτή σε αυτές τις περιοχές μπορεί να προβλεφθεί αποκλειστική πρόσβαση για τους αλληλείς εκείνης της περιοχής. Δεύτερη ερώτηση, συναφής. Ε, ποιο θα ήταν το κριτήριο για την επιλογή σκαφών και εξοπλισμών, αλλιευτικών εξοπλισμών που θα χρησιμοποιεί ο στόλος των αλλιών που θα έχουν την αποκλειστική πρόσβαση, διότι θα έλεγα ότι η αποκλειστική πρόσβαση σε συγκεκριμένε περιοχές για, για έναν περιφερειακό στολίσκο πρέπει να ε, υπακούει σε συγκεκριμένα κριτήρια για τα σκάφη και για τους εξοπλισμούς, ε, για την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, γι' αυτό το λόγο θα ήθελα, αν μπορεί η κυρία Ρόντο, να μας δώσει περισσότερε λεπτομέρειε. Ευχαριστούμε κυρία Πατρά, κυρία Φράγκα Ευχαριστώ. Εγώ δεν ε, ξέρω ακριβώ ποιε ήταν απόψει τη κυρία ε, Ρόντου, δεν είχα την ευκαιρία να την ακούσω. Δεν θα δώσω τη δική μου αλλά θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή. Βάσει και όσων είπε η Επίτροπος χθε ότι είχε προβλέψει ότι και στη Μεσόγειο να υπάρχει μια μέθοδος διαχείρισης, όπως έχουμε για τον Ατλαντικό, για τα υπόλοιπα κοινοτικά ύδατα έχοντας ε, κατά νου βέβαια ότι στη Μεσόγειο η μόνη ρύθμιση που υπάρχει είναι ο περίφημος κανονισμών τεχνικών μέτρων που ποτέ δεν έγινε σεβαστός ούτε προηγουμένως γιατί είναι αντιφατικός και παράλογος και ε, ούτε καν ε, τα αλληλευτικά εργαλεία δεν συνέπιπταν με τα ελάχιστα μεγέθη και τέλος πάντων δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Το θέμα είναι το εξή. Δεδομένου ότι στη Μεσόγειο τώρα δεν υπάρχουν τάκια ποσοστώσει με την εξαίρεση του ερυθρού τόνου, το σύστημα διαχείρισης ε, που υπάρχει στο βασικό κανονισμό και πάλι βασίζεται στι τάκια ποσοστώσει. Τα τάκια ποσοστώσεις δεν υπάρχει διαφορετικό μοντέλο δηλαδή από αυτό που έχουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αν στη Μεσόγειο σήμερα δεν έχουμε ένα μοντέλο που να βασίζεται σε τάκ και κότα, το μόνο μοντέλο διαχείρισης που μπορεί να είναι λογικό είναι η ελευτική προσπάθεια. Μοντέλο διαχείρισης μέσω της ελευτική προσπάθειας, το οποίο απορρίφθη από όλα τα κράτη-μέλη για την ε, γενική εφαρμογή, για να εφαρμοστεί γενικά στα κοινοτικά ύδατα. Έτσι λοιπόν, αν αυτό είναι το μοντέλο που θα εφαρμοστεί στη Μεσόγειο, αν πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει απορριφθεί για τα υπόλοιπα κοινοτικά είδατα, αυτό θα δημιουργούσε διάκριση. Εγώ πάντοτε ήμουν υπέρ του μοντέλου διαχείρισης έλεγχου της ελευθερικής προσπάθειας, γιατί νομίζω είναι το πιο εύκολο να ελέγξουμε και θα αποφεύγαμε κάθε πρόβλημα απορρίψεων, αλλά επειδή είναι ένα μοντέλο εύκολο να το λέξουμε, δεν το θέλει ούτε ο κλάδο ούτε τα κράτη-μέλη. Τώρα, βέβαια, αν κανεί δεν θέλει έλεγχο, ποιο θα είναι το μέλλον τη πολιτική, να το δούμε. Όμω, ε, αυτό που μου φαίνεται και απαράδεκτο είναι σε ένα μέρο των κοινωτικών υδάτων να εφαρμόζεται ένα σύστημα που θα βασίζεται σε ποσοστώσει και σε άλλο σε άλλη περιοχή όπως τη Μεσόγειο να χρησιμοποιείται ένα μοντέλο διαχείρισης ε, με βάση αλευτικής προσπάθειας. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις ιδέες που έχει η κυρία Επίτροπος, ε, τι βλέπει η Επιτροπή ως μέλλον, ε, να πούμε και εμείς τι μας αρέσει. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε θα έχουμε ένα μοντέλο διαχείρισης τη Μεσόγειο και να μιλάμε περί τίνο πρόκειται, γιατί το τάκι το μοντέλο τάκι ποσοστώσεων δεν θα ισχύει για τη Μεσόγειο. Τώρα η Κομισιόν α, θέλει να κάνει κάτι τέτοιο τη Μετσόγειο, αλλά εγώ θα ήθελα να είναι η Κομισιόν η πρώτη που θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Γιατί πράγματι ξεκινάμε από το μηδέν. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε, πριν να εκτεθώ εγώ, σε εκτεθεί η Κομισιόν που κάνει και τις προτάσεις. Και σε έρθει εδώ να μας τα καταθέσει. Και δεύτερον, για ε, να φέρω κάποια αντίρρηση σε εισαγωγικά στον κύριο Μελάνα. Εγώ είμαι υπέρ της και υπέρ ό,τι θέλετε, αλλά στη Μεσόγειο δεν είμαι υπέρ να έχουμε κατακαιρματισμό. Και θα σας πω το εξή κύριε Μιλάνα, εγώ είμαι εδώ πάρα πολύ χρόνια και έχω και πολύ πείρα. Και όταν εδώ κατατέθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτές τις ιδέες ότι είναι διαφορετική η Αδριατική, Προτάθηκε μια πρωτοβουλία και τέλος πάντων πουθενά δεν έφτασε, αλλά ήταν μια νομοθετική πρόταση Κομισιόν, ε, την εποχή της κυρίας Μολύν, όταν ε, λεγόταν ε, ότι δεν ο ε, και ο Μερλούκιος στην Αδριατική όπως στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Με τους επιστήμονες που μιλήσαμε μας είπαν ότι αυτό δεν ίσχυε και ότι οι στόλοι που έλειβαν εκεί απλώς ψάρευαν σε μια ζώνη συγκέντρωσης ηχθιδίων γιατί ε, δεν ήταν το πρόβλημα ότι αυτά τα είδη δεν μεγάλωναν στην Αδριατική αλλά απλώς ότι ελίευαν σε περιοχή με ηχθίδια. Εγώ λοιπόν ε, δεν θα διορούσα τη Μεσόγειο σε τμήματα, γιατί μπορεί να υπάρξει εισαγωγή διακρίσεων κατά των στόλων μας και αυτό θα είναι πολύ καλύτερο από το να έχουμε ε, ένα κανονισμό που να λαμβάνει υπόψη τα πολλαπλά είδη τα αλλιευμάτων ε, και τις ιδιαιτερότητες Μεσογείου και έχουμε και τα 12 μίλια, γι' αυτό έχουμε και τα διεθνή και τα όσα είπατε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το να δημιουργήσουμε κάποια κλειστά τμήματα στη Μεσόγειο, γιατί τελικά δεν είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα όσο πιστεύουμε και ε, εδώ να μην ακούγονται και διάφορες ιδέες, τους χαρή του Ομερλούκιος να μεγαλώνουν στην Αδριατική. Και έχω μια ερώτηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δούμε και αυτοί τι λένε, γιατί αυτοί καταθέτουν τις προτάσεις ε, στο θέμα αυτό και εμεί ε, στη βάση αυτή να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ή να τροποποιήσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως η Μεσόγειος όπως και η Βαλτική και όλες οι θάλασσες αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση. Δηλαδή κάθε θάλασσα έχει τα δικά της ε, γενή χαρακτηριστικά και αντίθετα με αυτά που μας έλεγε η Κάρμεν Φράγκα θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επανέλθουμε στις αρχές στις οποίες βασιστήκαμε στην αρχή της όλης διαδικασίας, μια ουσιαστική δηλαδή περιφερειοποίηση. Είναι προφανέ ότι στη Βόρεια Θάλασσα και στη Μεσόγειο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και άρα χρειαζόμαστε αυτή την ε, περιφερειακή προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως ε, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση αναλύευμα. Επίσης ε, να αποτιμούμε τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των προγραμμάτων, τις επιπτώσεις επί συγκεκριμένων ειδών, δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε για την Μεσόγειο όπως και παντού αλλού, στη Βαλτική, στη Βόρεια Θάλασσα κτλ. Χρειαζόμαστε ε, μία διαχείριση που θα βασίζεται σε αυτό το περίφημο κουτί εργαλείων και μία ουσιαστική περιφερειοποίηση. Ε, δεν ξέρω για αυτό το θέμα ποια είναι η θέση της Επιτροπή ε, και τη εισηγήτριας. η Κάρμεν μας το υπενθύμησε ότι στη Μεσόγειο δεν χρειάζεται, δεν υποχρεωτική διαχείριση των ελλειμμάτων βάσει των μεγίστων επιτροπών επιτρεπωμένων αλληλευμάτων, το ΤΑΞ ε, και όντω διαφέρει η κατάσταση στη Μεσόγειο σε σχέση με όλε τι υπόλοιπε. Δίκιο έχει, ε, Κάρμεν, αλλά η μοναδική μέθοδο που μπορούμε σήμερα να χρησιμοποιήσουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι να βασιστούμε στι αλληλευτικέ ε, προσπάθειε. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο βέλτιστο τρόπο διαχείριση των αποθεμάτων. Υπάρχουν βέβαια με πολλά κράτη-μέλη που αντίθεται σε αυτή τη μέθοδο. Θα μπορούσαμε επίση να ασχοληθούμε και να ρίξουμε το βάρο στην επιλεκτικότητα των εξοπλισμών ή στι κοινωνικέ κοινωνικό χώρο ταξικές ε, διαστάσεις ε, των αλλιευτικών ε, ζωνών και κάτι να προσθέσω διότι αυτό συνιστά πραγματική ιδιαιτερότητα για την Μεσόγειο. Όταν τα μεικτά αλλιεύματα μοιραζόμαστε με τρίτες χώρες όπως τη Μεσόγειο χρειαζόμαστε προφανώς εναρμονισμένους όρους σε διεθνές επίπεδο το οποίο δεν είναι καθόλου απλό στα πλαίσια των αρμόδιων οργανισμών εφαρμόζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα γιατί είναι καλή καλύτερα, πολύ και στι υπόλοιπε ε, θάλασσε, θα πρέπει σταδιακά ε, να ε, μειώνονται να μειώνεται η ελευθερική προσπάθεια και θα το επαναλάβω. Καλύτερα να επαναλαμβάνω κάποια πράγματα παρά να μην αναφέρονται καθόλου. Αυτό το σύστημα των μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία περίπτωση κατάλληλη για τη Μεσόγειο και για καμιά άλλη θάλασσα. Πρέπει να διατηρηθεί ο κοινωνικο-οικονομικός ιστός, ο οποίος θα καταστραφεί αν εμπορευματοποιήσουμε την πλεονάζουσα, την υπεραλίευση. Αν κατακλείδη, ε, ένα περιφερειακό σύστημα διαχείρισης είναι απαραίτητο ε, για την Μεσόγειο και Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε τα τεχνικά μέτρα αναλύευμα αλλά και όλα τα μέτρα που θα είναι προσαρμοσμένα ε, στη Μεσόγειο, στην βιομηχανία, ε, στην ε, συγγνώμη, αλία, την ερασιτεχνική μικρής κλίμακας γιατί αποτελεί μεγάλο ποσοστό στη Μεσόγειο. Και όλα αυτά τα προβλήματα και τι ιδιαιτερότητε που βλέπουμε σε άλλε θάλασσε είναι ακόμη πιο τονισμένε στη Μεσόγειο. Σα ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο ε, εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω ορισμένα από τα ζητήματα που ακούστηκαν στη ζήτηση σήμερα και να σκιαγραφίσω κάποιες απαντήσεις βασισμένες στην θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως την περιλάβαμε, τις περιλάβαμε μάλλον στην πρόταση που καταθέσαμε. Η Κομισιόν δεν προτείνει διαφορετική αλληλευτική πολιτική για την Μεσόγειο. Η μεταρρύθμιση έχει ως σκοπό να λάβει υπόψη τις διαφορετικές περιφερειακές καταστάσεις, διάφορες θαλάσσιες λεκάνες και εμείς προτείνουμε αλλαγή των ειδικών χαρακτηριστικών της Μεσογείου όπως αυτά ε, λαμβάνονται υπόψη στον κανονισμό της Μεσογείου. Ορισμένοι από εσά τονίσατε ότι πρέπει να λειτουργήσει ο κανονισμός για τη Μεσόγειο. Ασφαλώς αυτό θα αποτελέσει πρόκληση για τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν δηλαδή ώστε αυτό να υλοποιηθεί πράγματι. Η πρόταση που έχουμε καταθέσει για την περιφερειοποίηση, για παράδειγμα, βασίζεται σε ένα μοντέλο, διότι αυτό που καταθέσαμε είναι στην ουσία το μοντέλο το οποίο, στο οποίο βασίζεται ο, κανονισμός της Μεσογείου τώρα. Δηλαδή οι χώρες μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στα δικά τους ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αλληλείας αλλά και τις ε, θαλάσσιας δεκάνης. Νομίζω ότι το λάβουμε αυτό ως βάση για να ε, φτιάξουμε ένα ευρύτερο μοντέλο περιφερειοποίησης. Εμείς αυτό που προτείνουμε δεν είναι υποχρεωτικό μοντέλο, υποχρεωτικό το σύστημα. Δεν λέμε οπωσδήποτε πώ θα γίνει η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, διότι θέλουμε καλύτερα οι χώρε μέλη να αναπτύξουν τρόπου για να συνεργαστούν σε μια δεδομένη ε, θάλασσα. Ορισμένοι από εσά θέσατε το θέμα των τρίτων χωρών. Είναι ζήτημα κυρίω τη Μεσογείου, αλλά όχι μόνο. Συμβαίνει και σε άλλε ε, θαλάσσιες λεκάνε, αλλά για τη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχουμε επιτάπητο μια πρόταση που στοχεύει στην εξασφάλιση ότι θα γίνουμε εμεί ισχυρότεροι απέναντι στι χώρε αυτέ και θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα όλα τα εργαλεία που έχουμε στη θέση μα για να βελτιωθεί η συνεργασία και σε συμφωνία και στις συμφωνίες μάλλον με τρίτες χώρες να στοχεύουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας ώστε να λειτουργούμε ως ένα ενιαίο σύστημα σε κάθε θαλάσσια λεκάνη. Ανεξαρτήτως αν μιλούμε για χώρες Μεσογείου ή για τρίτες χώρες. Ασφαλώς πρώτοι εμείς πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα. Αυτό είναι ένα ε, από τα θεμελιώδη μηνύματα για να λειτουργήσει σωστά άλλωστε και ο κανονισμό τη Μεσογείου. Ο κ. Μιλάνα είπε προηγουμένω. και για τους ελέγχου, που είναι σημαντικό θέμα για τη Μεσόγειο. Για τα μέτρα διαχείριση έχουμε την ιδιαιτερότητα της Μεσογείου που σημαίνει δεν έχουμε ποσοστώσεις και τάκ για ορισμένα είδη. Η πρόταση δεν το αλλάζει αυτό. Δηλαδή εξετάζουμε πώς η διαχείριση της προσπάθειας θα γίνει πραγματική. Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη Μεσόγειο, να ξεφύγουμε από κάποια στοιχειώδη ε, ε, στοιχεία σχεδίων διαχείρισης που σημαίνει ότι διακόπτεται η αλληλεία για ένα μήνα ή δύο ας πούμε, να γίνουν πιο επιστημονικά τα σχέδια διαχείρισης, κάτι το οποίο είναι επιθυμητό και ε, αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί. Για τις απορρίψεις τώρα, που έχουν συζητηθεί πολύ τελευταία. Το θέμα είναι, ε, μάλλον οι απορρίψεις είναι θέμα και στη Μεσόγειο, που όπως είπα δεν έχει ποσοστώσεις και τάκ, αλλά έχουμε προβλήματα με τα ηχθίδια κλπ. Και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί είναι σημαντικό για την βιωσιμότητα των αλλιευμάτων. Βλέπετε στην πρότασή μας ότι λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση και ότι αυτή είναι περιπλοκότερη στη Μεσόγειο λόγω των διαφορετικών ειδών και αλίας και της αναμειξής τους. Θα χρειαστούμε λοιπόν και χρόνο, θα χρειαστούμε και πιλωτικά προγράμματα, θα χρειαστούμε και την στήριξη του ισχύοντος ταμείου, του, του νυν ταμείου αλλά και του μελλοντικού για να πετύχουμε μια καλύτερη επιλεξιμότητα για να μπορέσουμε έτσι μετά να αποφύγουμε τις απορρίψεις. Άκουσα και ανησυχίες σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστούν τα εχθήρια... στην υποχρέωση ε, να λαμβάνεται αυτό υπόψη όταν φτάνουν και εκφορτώνονται. Το βασικό μήνυμα πρέπει να είναι ότι οι χώρες μέλη είναι αυτές που δέχονται την πρόταση αυτή και θα πρέπει να είναι ικανές να καθιερώσουν κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τις καταστάσεις που ενδέχεται να ισχύουν σε ορισμένες χώρες μέλη, εκεί όπου δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, ε, εγκαταστάσεις μεταποίησης, όπου υπάρχουν ενδεχομένω παράλληλες αγορές και ούτω καθεξής. Αυτά είναι σημαντικά και θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή των εθνικών διοικήσεων για να μπορέσουν έτσι να υπάρξουν οι συνθήκες για να λειτουργήσουν καλά τα σχέδια διαχείρισης. Και το τελευταίο, τα TFC, γνωρίζουμε ποια είναι η πρόοδος της εφαρμογής των TFC. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το περιθώριο που αφήνουμε με την πρόταση στις χώρες μέλη να σχεδιάσουν ένα σύστημα που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της θαλάσσιας δεκάνης, τις ανάγκες των αλλιών τους και τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να λάβουν που τις έχουμε περιγράψει στην πρόταση γιατί θέλουμε οι χώρες μέλη να είναι σε θέση να καθιερώσουν τις προφυλάξεις εκείνες που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα της βιοτεχνικής αλίας, να μην υπάρχει δηλαδή έντονη κερδοσκοπία και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι είναι δυνατά αυτά, αλλά δεν θέλαμε να τα κάνουν κάθε υπαγόρευση. Άρα υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει, έτσι ώστε οι χώρες μέλη να εντοπίσουν ποια πράγματα θέλουν να προστατεύσουν ποια θέλουν να αποφύγουν και μετά εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους για να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα safeguard είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και ότι βέβαια θα αντέξουν και στην κρίση του δικαστηρίου ενδεχομένω. Ευχαριστώ κύριε Ροντούστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις και τους συναδέλφους που με παρακολούθησαν. Έχω την εντύπωση ότι διαμορφώνεται μια βασική συνένεση για τα όσα είπα. Η γεγονό είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε ώστε και η Μεσόγειος να μπορεί να παράγει καλύτερα και να εξασφαλίσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Φράγκα ότι ο οργανισμός για τη Μεσόγειο πρέπει να επανεξεταστεί. Είχε εκπονηθεί σε μια περίοδο όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε τη δυνατότητα να συμπράξη. Εξετάζοντας πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός τώρα, είπα προηγουμένως ότι πρόκειται για πραγματική καταστροφή και επιμένω στο χαρακτηρισμό αυτό. Αυτός ο κανονισμός είτε έχει, περιλαμβάνει, περιέχει δηλαδή σημαντικά σφάλματα ή τότε οι υπεύθυνε εθνικές κρατικές αρχές δεν ενδιαφέρονται, δεν εγκύπτουν επαρκώς στην εφαρμογή του. Αυτά πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Για την ερώτηση κ. Πατραονέβες έχω να πω το εξή. Είναι ιδέα πολλών από αυτούς που ανέφερα προηγουμένως, διότι εμείς εργαζόμαστε μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας εργασίας και διαρωτώμεθα αν είναι δυνατόν σε ορισμένους τομείς σε ορισμένου τομεί να ψαρεύονται ορισμένα μόνο ένα ή δύο ψάρια και να αναλαμβάνουν την ευθύνη οι ψαράδες. Και ίσω είναι και δυνατόν οι ψαράδες να παρακολουθούν οι μεν τους δε και να φροντίζουν με τον τρόπο αυτό να αποτρέπουν κάποιους να υπεραλλιεύουν. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και προτάσεις σχετικά από τις άλλες και τους άλλους συναδέλφους. Θα υπενθυμίσω και τη χθεσινοβραδινή συζήτηση με την Επίτροπο που είπε ότι το Συμβούλιο είπε εντάξει για τις απορρίψεις αυτό είναι σημαντικό και για τη Μεσόγειο, αλλά πρέπει να διατυπώσουμε ένα σαφή ορισμό. Εγώ νομίζω ότι ο ορισμός του ποιος είναι μικρός αλλιεύς ακόμα δεν έχει διατυπωθεί σωστά. Δεν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο το μήκος του σκάφους. Νομίζω μάλιστα ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Θυμηθείτε τα κινητά τηλέφωνα. Πριν από 5-6 χρόνια ακόμα ήταν διπλάσια και τριπλάσια σε μέγεθος από αυτά που είναι σήμερα. Βοηθήστε με λοιπόν στις προτάσεις να καταθέσετε και στις προτάσεις και να καταφέρουμε με κοινή προσπάθεια να τα φέρουμε σε αίσιο Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Ας ε, περάσουμε τώρα στο σημείο 10 η οργάνωση αγορών στον τομέα προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε δύο ανταλλαγές, υλοποιήσει δύο ανταλλαγές απόψεων στο παρελθόν. Στις 25 Ιανουαρίου κάναμε και μια κρόση για το θέμα αυτό. Και τώρα ο κύριος Στίβενσον θα μας παρουσιάσει το σχέδιο της έκθεσης. Ο κύριος Στίβενσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για την παρανόηση προηγουμένως. Όλοι έξω ήμασταν στις 10 και όπως σωστά είπατε μας ενημέρωσαν εσφαλμένο ότι θα αρχίζατε στις 10 και και πήγαμε για καφέ ε, αντί να έρθουμε στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας. Ε, όχι ότι το προτιμούμε, τέλος πάντων απ' έξω ήμασταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να, για να ξαναγίνει νέα συζήτηση για την έκθεση μου. Ούτως ή άλλως έχουμε κάνει ανταλλαγές απόψεων, έχουμε κάνει την προκατακτική συνεδρίαση επίσης ε, με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, τώρα έχω υποβάλει τροπολογίες ε, για το σχέδιο του κανονισμού που τροποποιούμε τώρα και θα ήθελα να σχολιάσω τις αρχές που διέπουν το σχέδιο. Πρώτον, δεν αναφέρονται στις γενικότερες προτάσεις της μεταρρύθμισης ε, ε που σχετίζονται με τις εμπορικές συναλλαγές. Εγώ πρότεινα για τις μελλοντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατηρηθεί αυτό το status quo στο μέτρο του δυνατού επειδή λειτουργεί εύρυθμα το σύστημα στη συνέχεια. Ο μελλοντικό ρόλο των οργανώσεων ε, παραγωγών, ε, κυρίω αν τροποποιηθούν τα σχέδια διαχείριση των αλλιευμάτων, θα πρέπει να υπακούει ε, σε συγκεκριμένα κριτήρια, παραδείγματο χάρη ο αριθμό των μελών κάθε ομάδα παραγωγών και άλλα σχετικά ζητήματα. Προτείνω όταν υπάρχουν ομοσπονδίε ενώσεις παραγωγών ή υπερεθνικέ ομάδε παραγωγών να ισχύουν κοινοί και δεσμευτικοί δεσμευτικοί κανόνε. Επίση, ε, κάνω διάφορε προτάσει για την επισήμανση. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρη ενημέρωση για του καταναλωτέ, ε, για την προέλευση, να ενημερωθούμε για τη μέθοδο παραγωγή και συλλογή των στατιστικών δεδομένων. να Αναφέρεται ο τρόπο αλλία με τρόπο που να αναγνωρίζει ο καταναλωτή. Επίση, η ημερομηνία εκφόρτωση πρέπει να είναι υποχρεωτική ε, και θελοντική θα είναι η αναφορά στην ημερομηνία αλλία. Ε, και ε, πάνω στην ε, ετικέτα μπορούμε να προσθέσουμε διάφορες άλλες πληροφορίες όπως βλέπετε στις προτάσεις μου. Αναφέρομαι δε και στο οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες όπως οι δοκιμές DNA ούτως ώστε να αποτραπούν η παραγωγή και να μην δίνουν σφαλμένες πληροφορίες προς τους καταναλωτές. Επίσης, υπάρχουν διάφορες δράσεις ε, για την χρησιμοποίηση ε, των ψαριών ε, για αγαθοεργίες. Πιστεύω ότι αυτό στρεβλώνει την αγορά. Τώρα σε σχέση με τις εκφορτώσεις, εφόσον ισχύει η απαγόρευση απορρίψεων, αν παρόλα αυτά εκφορτωθούν ακατάλληλα ψάρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τροφή ψαριών ή για την παραγωγή ηχθιελαίου και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καλύψουν τα ίδια το κόστος. Επίσης, ενθαρρύνω την χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλίας των νέων τεχνολογιών, ούτω ώστε να συνδυάσουμε πληροφορίε που ήδη είναι διαθέσιμες βάσει του VMS και των ηλεκτρονικών ημερολογίων απλοίου, ώστε να αυξήσουμε την κερδοφορία για ολόκληρο τον κλάδο. Επιπροσθέτως ε, προτείνω να ισχύσουν ε, οι εξαιρέσεις και ο κανονισμός από 1η πρώτου 2014 με αναθεώρηση να προβλέπεται ε, για το 2019 από τα τρία θεσμικά όργανα με πλησίασαν διάφορα μέρη της Επιτροπής που ζητούν επιμήκυνση της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογίων. Αρχικά είχε προβλεφθεί για την 20 29η Μαρτίου και ήταν ήδη παράταση. Η αρχική ημερομηνία ήταν 26 Μαρτίου και μετά την πρώτη παράταση και μετά τις πρωινές μας συζητήσεις θα ήθελα να προτείνω να εγκριθεί η 12η Απριλίου και μετα τις πρωινε νέα προθεσμία, 12 Απριλίου, εάν αυτό ικανοποιεί τα μέλη της Επιτροπής και έχετε όλοι επαρκή χρόνο για να προετοιμαστείτε εφόσον πρόκειται για σχέδιο νομοθετικής πρότασης και χρειαζόμαστε τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τέσσερα άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Καταρχήν η κυρία Λοβέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Στίβεν. Ε, ε, ήσουν εξαιρετικά περιεκτικός ε, στη παρουσίαση και στην έκθεσή σου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που φτάσαμε επιτέλους στην συζήτηση των τροπολογιών. Τις βλέπουμε γραπτός. Θα ήθελα να τις σχολιάσω. Λοιπόν, τροπολογία 1 Έχουμε ήδη συζητήσει αυτό το θέμα. Οι κανόνες του ΠΟΕ ε, και η όλη ιδέα ότι ε, θα πρέπει να ισχύσουν οι βιώσιμες αλληλευτικές πρακτικές και όλες οι σχετικές απαιτήσεις. Κοιτάξτε, για κάποιους αυτό κρύβει αντιφάσεις. Ε, όπως είδαμε και στην έκθεση Γκάλαχερ, και το πώς θα ε, γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα γίνουν δεκτά στον ΠΟΕ νομίζω ότι δείχνουν ε, ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή και ότι υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τροπολογία 3, εκεί που παραπέμπεται στην αιτιολογική σκέψη παριθμών 7 σχετικά με τον αριθμό των ε, ομάδων παραγωγών που υπάρχουν, ίσως αυτό είναι λεπτομέρεια όπως παραείμαστε συγκεκριμένοι για να αναφέρουμε κάτι τέτοιο σε κανονισμό, γιατί ούτως ή άλλως και αυτός ο κανονισμός κάποια στιγμή θα τροποποιηθεί. Τροπολογία 4, εδώ θα θέλετε να διευκρινίσετε ε, τον ελάχιστο αριθμό μελών ε, ως προς τα κριτήρια για την αναγνώριση, την καταχώρηση των ομάδων παραγωγών. Θα μπορούσατε ίσως να επεκταθείτε για αυτό το θέμα, ε, διότι δεν είμαι σίγουρη ε, τι ακριβώς καλύπτουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι χρειαζόμαστε ξεκάθαρα κριτήρια για τη σύσταση, αναγνώριση των ομάδων παραγωγών. Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένοι πρέπει να είμαστε και αν πρέπει να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένο αριθμό μελών της ομάδας ξέρω χρειάζεται. Ε, ας περάσω σε κάποια σημεία για τα οποία δεν συμφωνούμε, Στίβεν. Ε, πρώτον, ε, η ανάπτυξη αυτού του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ecolabel. Έχω την ε, εντύπωση ότι είναι θετικό να έχουμε ελάχιστα κοινά πρότυπα για οποιοδήποτε οικολογικό σήμα Υπάρχουν ε, ήδη ε, διάφορες ε, προτάσεις για αναθεώρηση για τα όσα ισχύουν για τα οικολογικά σήματα που ενδεχομένως να γίνονταν και αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως δεν θεωρούμε ότι η Επιτροπή ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβουν αυτό το ρόλο του πιστοποιητή ενός οικολογικού σήματος. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή θα ταυτίζεται με ένα οικολογικό σήμα γιατί τα συγχαίουμε αυτά τα δύο. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς ρόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει ε, πόσο μπορούμε να ξεπεράσουμε ε, τους κανόνες ως προς το, το οικοσύμα δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποια ιδιότητα, ποιο ρόλο θέλουμε να προσδώσουμε στην Ένωση σε σχέση με το σήμα ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Τα ίδια είχαν γίνει ε, και πριν από λίγα χρόνια είχαμε αυτό το θέμα της κλίμακας από το Α μέχρι το σιγμα τάφη για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα για τα ψυγεία και στη συνέχεια είχαμε κάποια ψυγεία που είχαν την χαμηλότερη βαθμολογία ε, F σίγμα τάφε και οι καταναλωτές πήγαιναν αυτόματα να πάρουν τα ψυγεία με βαθμό ε, Α και σήμερα όλα τα ψυγεία είναι α στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς, κανείς δεν θέλει να χάσει το α του και τώρα βγάλαν καινούρια α συν, αλφα συν συν, συν συν συν και όλες τις σχετικές ε, βαθμολογίες. Ε, να, σε αυτή την κατάσταση θα περιέλθουμε στην Ένωση αν προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε δικό μας ε, οικοσύμα. Κάποιοι μου είπαν ότι θέλουν να εισαγάγουν και κοινωνικά κριτήρια μέσα στο οικοσύμα. Τι θα έχουμε στο τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εγγυάται τα υψηλά ε, ποιοτικά πρότυπα, οποιαδήποτε πρότυπα, είτε είναι οικολογικά είτε είναι κοινωνικά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχω ένα πρόβλημα με τα οικοσύματα και δεν θέλω να έχουμε τέτοια ε, ψεύτικα ψευδοοικοσύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε κριτήρια για τα σήματα, αλλά ποιο είναι ο ρόλος αυτών των σημάτων να προωθήσουν την ανάπτυξη, ούτω ώστε στη συνέχεια την επόμενη χρονιά να αναθεωρήσετε τα κριτήρια και να γίνετε αυστηρότεροι για τα περιβαλλοντικά κριτήρια ή τα κριτήρια ως προς την ευημερία των ζώων ή οποιαδήποτε κριτήρια. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, ο κίνδυνο είναι να ε, διατηρηθεί όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε με άλλα σήματα και το αποτέλεσμα θα είναι να χαμηλώσουν ε, τα πρότυπα. Ε, διότι όλοι προσπαθούν, θα προσπαθήσουν ε, να κερδίσουν κάτι από αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσδώσουμε αυτό το ρόλο του πιστοποιητή των σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Λεβίν, μπορείτε σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε, λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρο, θα ήθελα, επιτρέψτε μου, να προσθέσω κάτι τελευταίο. Δεν έχουμε χρόνο. Ένα τελευταίο. Για την τροπολογία 11 διαγράψατε την επεξεργασία των ανεπιθυμήτων αλλιευμάτων ε, από τους στόχους των ομάδων ε, παραγωγών. Ε, μπορείτε να επεκταθείτε για ποιο λόγο ακριβώς το κάνατε. Κατόπιν ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ε, τροπολογία 18 Στρούεν άλλαξε το ποσοστό του 40% για τους παραγωγούς υδατοκαλλιεργείων και τώρα είναι 65% αυξήθηκε. Ε, γιατί η Επιτροπή προτείνει όμω 40% και όχι 65% θα μπορούσες να μου το εξηγήσει. θα σου ήμουν ευγνώμων. Τέλο, τροπολογία 21. Ε, προτείνεις ε, οι ομάδες ε, παραγωγών να συγχρηματοδοτούν και μόνο την αποθήκευση των προϊόντων. Η Επιτροπή προτείνει να χρηματοδοτούν, όχι να συγχρηματοδοτούν οι παραγωγοί. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, από τους τέσσερις που είχαν ζητήσει το λόγο, τώρα περάσαμε στους οκτώ. Θα δώσω και στους οκτώ το λόγο, αλλά σας παρακαλώ τρία λεπτά. Θα σας περιορίσω στα τρία λεπτά. Ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα οργανωθώ για να μου κόψετε το μικρόφωνο. Καταρχήν ευχαριστώ Στρούαν που μας έδωσε ε, και άλλη προθεσμία για τις ε, τροπολογίες, ε, αν και είχαμε εργαστεί για να τις καταθέσουμε στις 26. Και να σε ευχαριστήσω για την έκθεση που είναι εξαιρετικής ποιότητας. Γενικά οι τροπολογίες του συγητή με βρίσκουν σύμφωνο. Βέβαια υπάρχουν ε, κάποια σημεία που πρέπει να συμπληρωθούν, να προσθεθούν, ε, διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα. Σκέφτομαι τη σημασία τη προσαρμογή ε, τη εμπορική και τελωνική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη κοινή πολιτική. Καταρχήν, για να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των εισαγωγών προϊόντων, όλοι συμφωνούμε με αυτό, για την αρχή τη αμοιβαιότητα, ε, να ε, έχουμε αυτή την αρχή στα πλαίσια των διμερών και πολυμερών συναλλαγών και επίση βάση ενό δίκαιου ανταγωνισμού. Ιζαμπέλα, το συζητήσαμε αυτό μόλις, το δεύτερο σημείο, είμαστε υπέρ και το υπογραμμίσαμε σε προηγούμενη έκθεση. Η κυρία Φράγκα επίση το έχει κάνει πριν από μένα. Δημιουργία ενό ε, Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματο. Η Κομισιόν πρέπει να καταθέσει μια πρόταση κανονισμού για να δημιουργηθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα που θα πρέπει να παρουσιαστεί στους νομοθέτες μέχρι την 1η, 1η 2015. Κατά την άποψή μου ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, υπάρχουν πολλά εμπόδια, αλλά είναι απαραίτητο σήμερα και πρέπει να καθορίσουμε ε, αυτό το σήμα για να είναι στο δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Κατόπιν, οργανώσει παραγωγών πολλές φορές ε, θέτουν κάποια μέτρα διαχείριση ορισμένων λευμάτων πέραν αυτών που προτείνει η Κομισιόν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του αφήσουμε αυτή τη ε, δυνατότητα, γιατί πηγαίνουν ακόμα παραπέρα και μου φαίνεται ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τις Στρούαν, το ανέφερες προλίγου. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και για μη διατροφικού σκοπούς, μη επιστημονικούς σκοπού και όχι μόνο δίνουν σε φιλανθρωπικέ για όλα αυτά τα σημεία, αλλά για αυτά θα σου προτείνω κάποιες τροπολογίες. Αλλά συνολικά είναι πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική και μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Τρία λεπτά. Θα βάλω το δυνατά μου για ένα σε χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Στρούαν. Νομίζω ότι η έκθεση μας παρουσίασες είναι πολύ καλή. Γιατί η προστασία του καταναλωτή είναι το κύριο στοιχείο που προκύπτει από την εκθεσή σου. Δεύτερον, ε, ανταγωνισμός, ε, αλλά δίκαιος και ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός σε μια αγορά που είναι η μεγαλύτερη αγορά λευτικών προϊόντων και προϊόντων καλλιέργεια σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό μου φαίνεται τόσο σημαντικό τα κριτήρια να είναι ταυτόσιμα για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή. Οι οργανώσει μα παραγωγών πρέπει φυσικά να είναι αυστηρέ και να υποβάλλονται στα πιο ψηλά κριτήρια ποιότητα. Πολύ ωραία, αλλά το, πρέπει, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τα εισαγόμενα προϊόντα και αυτό αφορά και τον ΠΟΕ και συγγνώμη, την ΚΟΑ και το ε, συζητήσαμε σε περίπτωση παραδείγματος χάρη του Παγκάσιου. Ε, μπορεί πολλές φορές ε, αυτό το ψάρι να περιέχει βαρέα μέταλλα, το έχουμε συζητήσει. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το μελετήσουμε εις βάθος, σε ό,τι αφορά τώρα τα περιπίπτοντα λιεύματα. Και αυτό που θα πρέπει να εκφορτώνουμε στο μέλλον. Να μπορούν αυτά τα ψάρια να μετατραπούν σε αλεύρα που να συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Όπως ε, είπα, εμείς ως ε, μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά πρέπει να παγιώσουμε τη δική μας ήχθιο και δεν το καλλιέργεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της ΚΑΛΠ όταν μιλάμε για χρηματοδότηση πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά βέβαια αυτό κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που θέλω να τονίσω εγώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούνη, κυρία Φράγκ. Ευχαριστώ. Εγώ θα αναφερθώ γρήγορα στις ε, τροπολογίες, Να σας πω ότι είμαι υπέρ της οικολογικής ετικέτας ε, και πέρα ε, των δισταγμών ε, της κ. Λοβέν, ε, αν ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΦΑΟ δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να εφευρούμε τίποτα το καινούριο. Δεύτερον, για να δούμε τις τροπολογίες. Στις τροπολογίες 11 και 13, επί της αρχής δεν συμφωνώ. Αυτό, όπω είδατε από... Ε, αυτό έχει να κάνει και με την απόφαση που θα πάρουμε για τι απορρίψει. Αν πάρουμε κάποια απόφαση σχετικά με αυτό, κάποιο θα πρέπει να το κάνει. Αυτό εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού δύο τροπολογιών. Στην τροπολογία 16 εγώ πέρα από τη διαγραφή θα ήθελα να μου εξηγήσει η Επιτροπή τι εννοεί με αυτή τη δεσπόζουσα θέση. Γιατί αυτό πρέπει να μας ε, ξεκαθαρίσει. Στην 18 η Κομισιόν ε, θα ήθελα να μου δικαιολογήσει το 40% γιατί ε, δεν έχουμε το ίδιο ποσοστό για την ιδιωτοκαλλιέργεια και για την αλία. Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι το ίδιο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν έβαλε το 40%. Στην περίπτωση της τροπολογίας 21 δεν συμφωνώ με τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση. Θα πρότεινα να έχουμε τον όρο χρηματοδότηση όπως την ε, πρόταση της Κομισιόν στην τροπολογία 22. Η ευελιξία που θέλετε να δώσετε εδώ είναι υπερβολική. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο οι οργανώσεις παραγωγούν πριν να ξεκινήσει η περίοδος να κάνουν την πρόταση, γιατί στην πρότασή τους ε, μπορεί να οδηγήσει σε κάποια μπερδέματα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τώρα την 23, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτό που λέει η πρόταση της Κομισιόν και αυτό που λέτε εσείς. Δεν νομίζω ότι το ένα αποκλεί το άλλο. Για την οικολογική ετικέτα το είπαμε. Ας περάσουμε λοιπόν ε, στην επισήμανση, στην 26. Εγώ θα πρότεινα όταν έχει ξεπαγώσει για να απολυθεί νοπό. Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διάκριση για την οπή πώληση. Γιατί αν χρησιμοποιηθεί το προϊόν συνέχεια για κονσέρβα δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για το 42.2 άρθρο θα έπρεπε ε, να διαγράψουμε ε, τα, ε, το 1604 και το 1605 ε, αυτές τις μερίδες γιατί προέρχονται από διαφορετικά μέρη αλίευσης και μπορεί τελικά να έχουμε τικέτες που θα είναι εντελώ δυσνόητες ή ακατανόητες και περνώ στην τροπολογία 29 για την εκούσια ενημέρωση τις πληροφορίες. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι ακούσεις πληροφορίες θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι θα πρέπει να μπορούν να επαληθεύονται. Πολύ ωραία να δίνονται αυτές οι πληροφορίες εκούσιοι, αλλά θα πρέπει να επαληθεύονται οι πληροφορίες αυτές. Δεν ε, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε εκεί οτιδήποτε. Να μπορούν να επαληθεύονται λοιπόν αυτές οι πληροφορίες. Πρέπει να το προσθέσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Φράγκα. Κύριε Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περάσω απευθείας στις παρατηρήσεις για να μην χάνω χρόνο. Θα ήθελα να κάνω την ίδια διάκριση με την κυρία Φράγκα ε, για την 18 πραγματικά, ε, ε, τροπολογία εννοώ 18, δεν καταλαβαίνω ούτε το ποσοστό του 40% ούτε την αλλαγή που έγινε ε, και την αύξηση σε 65% και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε παρακαλώ επίσης για τα παραρτήματα όπου αναφέρονται προϊόντα κονσερβοποιημένα με ε, διάφορα συστατικά από διάφορα λιεύματα ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να επανεξετάσουμε ε, αυτό τον κατάλογο για την όλη κατάσταση γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν αναφερόμαστε τώρα στην επιστημονική ονομασία του κάθε είδους, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος με τα γέννη των ψαριών διότι καλύπτονται πολλά διαφορετικά υποείδη και πιστεύω ότι αν γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου ε, θα ε, εξοικονομήσει πόρους ε, και ο ίδιος ο κλάδος. Θα ήθελα τώρα να θέσω και άλλα δύο κατ' εμέ πολύ σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, η ημερομηνία αλίεσε των αλλιευτικών προϊόντων ή των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας έχω την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί μια ε, παρανόηση. Όντως πρέπει να υπάρχει ασφάλεια αλλά δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τη σωστή ενημέρωση του ε, καταναλωτή. Δημιουργούνται αμφισημίες. Θα σας εξηγήσω. Όταν μιλάμε για ημερομηνία άλλη θα καταλάβει ο καταναλωτής ε, ότι πρέπει να αγοράσει το προϊόν που έχει την πιο πρόσφατη ημερομηνία. Όμως η ποιότητα είναι ε, σε άμεση συνάρτηση με την ε, μέθοδο ε, αλίας και δεν σχετίζεται μόνο με την ημερομηνία. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να δημιουργηθούν αμφισημίες. Το ίδιο για τα κατεψυγμένα προϊόντα. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει έλεγχος της ημερομηνία κατάψυξης, κυρίως όταν μιλάμε για εισαγόμενα προϊόντα και γι' αυτό θα θέλαμε να θεσπίσουμε ε, ε, προποθέσει τόσο ώστε να καταργηθεί αυτό ο αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα σε νόπα και κατεψυγμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρε ε, και μπορεί να φέρνουν ημερομηνία που εμεί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ελέγξουμε και άρα δημιουργούνται στρεβλώσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Τελευταία, α και το αναφέρω αυτό, διότι Μιλούσατε για την αναφορά στην ε, ημερομηνία αλίας ε, για τα ε, αλλιευτικά προϊόντα ή τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Τώρα, τελευταία ερώτηση σε σχέση με το οικοσύμα. Είμαι υπέρ χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια οντότητα, ποιος οργανισμός ε, θα αναλάβει την πιστοποίηση του ε, σήματος. Πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ε, και όχι οργανισμός του ιδιωτικού τομέα, διότι αναπόφευκτα θα πλεονεκτούν οι πελάτες αυτού του οργανισμού και το σήμα αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυπτεί όχι μόνο τα προϊόντα της Ένωσης, αλλά ε, και τα εισαγόμενα προϊόντα. Ας αλλάξουμε το χρώμα πάνω στο σήμα τουλάχιστον ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει ε, ποια ψάρια έχουν αλλιευθεί στην Ένωση και ποια είναι εισαγόμενα. Σας ευχαριστούμε κυρία Πατράου. Τρία λεπτά ο κύριο ε, Φερέιρα. Θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικός. Δεν προλαβαίνω σε τρία λεπτά να πω πολλά πράγματα. Ε, καταγράφουμε τις ε, προτάσεις ε, του κυρίου Στίβενσον και σε πρώτη ανάγνωση θα συμφωνήσουμε με κάποιες από αυτές, διαφωνούμε με άλλες, πάντως η γενικότερη αξιολόγηση είναι ότι είναι ανεπαρκής οι προτάσεις αυτές. Ε, είμαι η εισηγητής ε, της έκθεσης Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και μέσα στην έκθεση έχω μια ολόκληρη δέσμη προτάσεων που θα μπορούσατε και εσείς να συμπληρώσετε και να βελτιώσετε έτσι την πρόταση που τώρα εξετάζουμε. Πρώτο θέμα είναι σημασία να είναι ξεκάθαρες οι αρχές που εφαρμόζονται και αυτό δυστυχώ λείπει από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΚΟΑ, η Κοινή Οργάνωση Αγορά, έχει ω στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών και τη ε, σωστή ε, απόδοση ε, ω προ του παραγωγού, είτε μιλάμε για αλλιεύματα είτε για προϊόντα καλλιέργεια. Δεύτερον, βασίζεται αυτή η πρόταση σε μια πολύ σημαντική δομή, δηλαδή τι ομάδε παραγωγών. Όμω, είναι πάρα πολύ διαφορετική η κατάσταση ανακράτω ω προ την ανάπτυξη των εγχωρίων ε, ομάδων παραγωγών. Το αναγνωρίζει ο εισηγητή ε, και υπάρχουν μέτρα που όντω ε, θα πρέπει να υιοθετηθούν, αλλά θα πρέπει αυτό να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών για να λάβουν υπόψη τι ιδιαιτερότητε και το επίπεδο ανάπτυξη των εγχώριων ομάδων παραγωγών. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε εδώ τιμέ που θα αναγνωρίζονται για κάθε ομάδα παραγωγών χωρίς να αφήνουμε τον Εθνικό Αρμόδιο Οργανισμό να αποφασίζει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε δεόντως υπόψη ε, τις μεγάλες, ε, πραγματικά πολύ μεγάλες διαφορές ε, ως προς τις ομάδες παραγωγών ανακράτω μέλο μέλος. Στη συνέχεια ε, ε, Σα είπα ήδη ότι συμφωνώ με πολλέ προτάσει του κυρίου Στίβενσον, όπω παραδείγματο χάρη η πρόταση που κάνει για την ε, συμμετοχή ω προ την ενημέρωση των ομάδων παραγωγών για τα στατιστικά δεδομένα, για την κατάσταση των αποθεμάτων κτλ. Επίση, θα πρέπει να προβλέψουμε οικονομικά αντισταθμίσματα ελάχιστα που θα το επιτρέψουν στου παραγωγεί να καλύψουν το κόστο τη εκφόρτωση των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να προβλέψουμε οικονομική αντιστάθμιση ε, για να συνοδεύσουμε οποιαδήποτε πολιτική απαγόρευση των απορρίψεων. Πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί αυτό το κόστος ε, που ε, υφίστανται η παραγωγή κατά την εκφόρτωση αυτών των αλλιευμάτων στη συνέχεια. Αναφέρεστε στις σημερινές και θα κλείσω, το ξέρω ότι πέρασαν τα τρία λεπτά. Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, πολύ μεγάλε στρεβλώσει ω προ την προσθέμενη αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Ε, ε, υπάρχουν μεγάλες ε, ανισότητες ω προς την προστιθέμενη αξία και όσοι βρίσκονται κάτω-κάτω στην αλυσίδα ε, παίρνουν ένα ελάχιστο μερίδιο, δηλαδή η τιμή της πρώτης αγοράς θα πρέπει να αναθεωρηθεί ούτω ώστε σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού να μοιράζεται το κέρδος ισότιμα. Χρειάζεται δηλαδή να έχουμε ένα περιθώριο ελιγμών σε επίπεδο κράτους μέλους, ούτως ώστε ο αρμόδιος αργονισμός ε, να κάνει την αξιολόγηση, να λαμβάνει υπόψη την αρχική τιμή ε, πώληση, ε, την τελική τιμή του καταναλώτη και να γίνει ισότιμη κατανομή. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, είναι κατά βάση καλέ οι προτάσει της Κομισιόν. Και αυτά που προτείνει ο Στρούαν ξεκαθαρίζει, ξεκαθαρίζουν μάλλον και συμπληρώνουν τις προτάσεις αυτές. Με τον γενικό στόχο που έχουμε, δηλαδή μια κοινή οργάνωση αγοράς. Για τις τροπολογίες, για τα εκτιμώντας πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα ψάρια που έρχονται από τρίτες χώρες να ανταποκρίνονται στις ψηλές προδιαγραφές που διαθέτουμε. Για, τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες αιτιολογικές σκέψεις θεωρώ όντως ότι στη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική οι οργανώσει παραγωγών πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Δεν συμφωνώ τον κ. Φερέιρα ότι πρέπει να επιτρέψουμε στις χώρες μέλη να ρυθμίζουν οι ίδιες των ε, οργανώσεων παραγωγών που σημαίνουν διαφορετικά πράγματα οι διάφορες χώρες θα πρέπει να πούμε ακριβώ τι είναι οργάνωση παραγωγών, εφόσον μάλιστα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Μιλούμε για κοινή αγορά και μέσα σε αυτήν την κοινή αγορά χρειάζεται να έχουμε κοινά πρότυπα. Και αυτά προσπαθεί να επιτύχει ο Στρούαν Στίβενσον. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 3 των ε, αιτιολογικών σκέψεων, λέει τρει χώρε. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία να μπει μέσα και η Ιρλανδία και ίσως και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τροπολογία 6, αυτή, λέει ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν σαφείς πληροφορίες για τις ημερομηνίε και τη μέθοδο ε, αλλά πρέπει να γίνει πιο σαφή, διότι μιλούμε εδώ για διαφάνεια και ηχνητασιμότητα. Για την τροπολογία 18, θα έλεγα ακόμη περισσότερο. Πού το βρήκε το 42% η Κομισιόν και ο εισηγητής λέει 65%, εγώ θα έλεγα μάλιστα 85% και η τροπολογία 20% σε περίπτωση μη συμμόρφωση μπορεί να αρθεί η έγκριση. Εγώ μάλιστα θα έλεγα όχι μπορεί, όχι δυνητικά, όχι may, αλλά shall, θα αφαιρείται. Και μάλιστα άμεσα. Για την 21, αυτή η ερώτηση ήδη έχει τεθεί σχετικά με την συγχρηματοδότηση. Μιλούμε, όταν μιλούμε για συγχρηματοδότηση, μιλούμε για χρηματοδότηση που δίνεται και από τη χώρα μέλος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς εννοεί εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συγχρηματοδότηση και η τροπολία... Η ε, τροπολογία 23 Εδώ χρειαζόμαστε κίνητρα και αντικίνητρα. Θα πρέπει να δίνεται κάποια χρηματική αντιστάθμιση. Και για την 27 να καταστρώσει τις βασικές γραμμές η Κομισιόν και να βάλουμε και μια προθεσμία κοντά στο 2015 για να εφαρμοστεί η διάταξη για αυτή την επισήμανση. Αυτά που λέει η Λόβιν είναι σωστά. Αλλά για αυτή την οικολογική επισήμανση υπάρχουν επιχειρήσεις που δίνουν τέτοια σήματα οικολογικής επισήμανσης και που είναι στην πραγματικότητα απάτη. Thank um, Ευχαριστώ. Λίγα σχόλια πρώτα για την προθεσμία των τροπολογιών. Ο κ. Στίβενσον δέχεται παράταση μέχρι τις 12 Τετάρτου. Ο εισηγητής έχει δώσει επαρκή δυνατότητα και στους κ. εισηγητές να συζητήσουν μαζί του. Παρ' όλα αυτά Νομίζω ότι λίγο περισσότερο, λίγο μακρότερο χρονικό διάστημα της τροπολογίας θα διευκολύνει πολλούς για την επισήμανση και την εκφόρτωση και την ε, αλίευση κλπ. Νομίζω κατ' επιλογή θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία αλίευσης γιατί και οι καταναλωτές και οι έμποροι θα ωφεληθούν εάν γνωρίζουν ότι το ψάρι που αγοράζουν είναι όσο γίνεται πιο φρέσκο. Άλλο είναι το ψάρι που ψαρεύτηκε πριν από δύο μέρες, άλλο πριν από πέντε και άλλο πριν από μια εβδομάδα. Δεν είναι άσχημη ιδέα λοιπόν αυτή που προτείνει ο κ. Στίβενσον και η εκφόρτωση και στην ξηρά δηλαδή είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτή ότι η αλίευση έχει γίνει σε ένα τόπο που έχει καλή φήμη. και που εγγυάται και, την, και το, ψάρι είναι φρέσκο. Και οι καταναλωτές θέλουν ψάρια από ε, χώρες που έχουν καλό ιστορικό και για την οικολογική επισήμανση, το eco-labeling, ισχύει το ίδιο. Και εγώ προσωπικά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένη η διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η δε κομισιόν θα πρέπει να είναι η απότατη αρχή για αυτό το eco-labeling. Αν και εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι η υπατή αρχή για όλα τα πράγματα. Γιατί αυτό οδηγεί και σε πολλά μειονεκτήματα. Για τα παράλληλα, τα παρελκόμενα αλλιεύματα, και την κατάργησή τους, με, προσπαθώντας να λύσουμε το πρόβλημα των απορρίψεων, θα παρακαλέσω τον κύριο Στίβενσον να διευκρινίσει το περιεχόμενο της τροπολογίας 23 και είμαι και κάπως διστακτικός όσον αφορά το οτιδήποτε άλλο που μπορεί να θεωρηθεί παρελκόμενο αλίευμα να πάει να γίνει ηχθιάλευρο δηλαδή. Δεν είμαι βέβαιος αν η διατύπωση αυτή είναι αρκετά εύκαμπτη ώστε να αποφεύγεται η τέτοια κακή χρήση καλών κατά τα άλλα ψαριών. Μιράντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην πρόταση μεταρρύθμισης της ε, ΚΟΑ μας ε, λείπει και από το βασικό κανονισμό και από το γραφό εργασίας ε, η αναφορά και προσανατολισμός ε, έναντι του στόλου μικρής κλίμακας. Από πολλά μέτωπα που εργάζονται στον κλάδο της μικρής αλίας, της ρεστινικής αλίας, επέμειναν και άλλες οργανώσεις πέρα των οργανώσεων παραγωγών να αναγνωριστούν. Δηλαδή, να έχουμε μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση από αυτή που προτείνει η ίδια η Κομισιόν. Για να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για φόρο αλία, είναι απαραίτητο ο μεγαλύτερο προστατευτισμό από την πλευρά των δικήσεων. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά γιατί δεν αναφέρεστε στι προστατευόμενε ονομασίε προέλευση. Στην Γαλλικία έχουμε για ε, τα μύδια και ε, προέρχονται από έχουμε εγγύηση ποιότητας, ε, εγγύηση προέλευσης και μερικές φορές ε, ξέρετε ότι έχουμε και προϊόντα εισαγόμενα που δεν ε, σέβονται ε, τους ίδιους όρους, παραδείγματος χάρη προϊόντα που έρχονται από τη χιλή στην περίπτωση αυτή και στο στην τραπολογία 14 ε, ο εισηγητής ε, λέει ότι ε, θα πρέπει να προωθηθούν οι βιώσιμες δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία των Ελλήνων με τις τοπικές αρχές θα πρέπει να δούμε τι εννοούμε με τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια εκτατική ή εντατική. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Γέρο. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Στιβένσον για την έκθεση. Είναι η πρώτη μου δουλειά ως σκιώδης ε, και νομίζω ότι το έγγραφο του κ. Στίβενσον είναι πολύ καλό, το οποίο μας επιτρέπει να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να έχουμε και κάποια σημεία αφετηρίας για να εργαστούμε. Η ΚΟΑ είναι μία από τους κύριους, ένας από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης ε, πολιτικής και ξέρετε ότι εγώ συμφωνώ και ότι πρέπει να σεβαστούμε τους καθολικούς στόχους της μεταρρύθμισης ε, πολύ συγκεκριμένα και προς αυτή την κατεύθυνση μέσω αυτής της θητείας θέλουμε να βελτιώσουμε την θέση της ευρωπαϊκής αγοράς, να ενισχύσουμε τη δυναμικότητά μας ε, και να ενισχύσουμε τα προϊόντα έναντι των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα πολύ γρήγορα ρύθμιση της αγοράς ε, πρέπει να έχει μεταξύ των στόχων της και μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή και πρέπει να ηγηθούμε την μέγιστη δυνατή ενχνευσιμότητα μέχρι δηλαδή να γνωρίζει ο καταναλωτής όλη τη διαδρομή του προϊόντος από τη θάλασσα μέχρι το τραπέζι και να προσπαθήσουμε να παγιώσουμε και να βελτιώσουμε τη θέση μας ως Ευρωπαίοι έναντι του διεθνούς εμπορίου. Επίσης είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να αποφύγουμε και τον ντάμπικ από τις τρίτες χώρες. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να καθορίσουμε κάποιους κανόνες που μου ε, θα μας ευνοούν και θα μας αντιστοιχούν να ε, προσφέρουμε προϊόντα πρώτης ποιότητας ε, σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις παραγωγών και είναι και αυτές σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να έχουμε τις οργανώσεις παραγωγών αλλά και όλους τους ενδιαφερμένους στον τομέα επίσης πρέπει να μπορούν οι οργανώσεις που καλύπτουν μια μεγαλύτερη γκάμα από τον τομέα της αλίας μέχρι και την ερασταχνική αλία να μπορούν να είναι παρούσες και να δίνονται ενισχύσει. Είναι θεμελιώδες να προωθήσουμε τα προϊόντα έτσι ώστε το τομέας, ο κλάδος να γνωρίζει ε, ποια είναι ακριβώς η ποιότητα. Γι' αυτό πρέπει να διατηρήσουμε την ημερομηνία αλίευσης και την ε, οικολογική ετικέτα όπου θα γνωστοποιείτε πώς, με ποιο τρόπο έχουν ελευθεί και ποια είναι ε, η διατροφική ποιότητα του προϊόντος. Γιατί αναφερθήκατε σε κάποια ποσοστά, 80 ή 60%. Ε, για το 60% των προϊόντων που καταναλώνουμε δεν υπάρχει εγγύηση ποιότητα σε αυτά. Και ε, εμείς ε, θέλουμε να προστατεύσουμε ε, την ποιότητα και την ποικιλομορφία που προσφέρει το σύνολο της Ιβερικής Κερσονήσου στους καταναλωτές. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και με την ομοθεσία σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα είδη και τα ελάχιστα με συγχωρείτε μεγέθη και πρέπει να περιμένουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής και για τη βιώσιμη ελεία, για τη διατήρηση των πόρων, της θάλασσας, αλλά και την κοινωνική και οικονομική διάσταση και αυτά αποτελούν βάση του ορώματο μας από τη Σοσιαλιστική Ομάδα για το μέλλον της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ε, απαιτούμε η μελλοντική πολιτική της ΚΑΛΠ να διασφαλίζει την εφορία της Ελίας ε, και να διασφαλίσουμε και αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς διατηρώντας τις εργασίας και συνεισφέροντας όπως κάναμε μέχρι τώρα στο να διατηρήσουμε τον πληθυσμό στις παράκτητες περιοχές. Θα πρέπει να σεβόμαστε την ε, διατήρηση των οικολογικών συστημάτων, να σεβόμαστε τη βιοπικιλότητα, χωρίς να ξεχνάμε το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική και η οικονομική λειτουργία της Ελίας. Απλώς να πω ότι θα παρουσιάσουμε κάποιες παρατηρήσεις των συγητή, δυνάμει και με ακούστηκαν εδώ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ γρήγορα, κύριος Ντέβιτ. Θα είμαι σύντομος ε, και θέλω να υποστηρίξω πολλές από τις προτάσεις του Στρούαν, αλλά θέλω να τονίσω δύο θέματα που διαφωνώ. Καταρχήν, η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ε, παράγει η ίδια το οικολογικό σήμα. Αυτό είναι τρέλα. Έχουμε πάρα πολλέ οικολογικέ ετικέτε, ε, όπω έχουμε από το Συμβούλιο Επιστασία ε, των Θαλασσών, παραδείγματο χάρη. Προτάθηκαν και άλλε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θέτουμε κριτήρια για τη χρήση των ετικετών στα προϊόντα, αλλά το να το κάνουμε εμεί οι νομίζω ότι όχι απλώ θα υπάρχει επικάλυψη φυστάμενε προσπάθειε και δεν θα δημιουργηθούν και προβλήματα που θα είναι δύσκολο να λύσουμε, αλλά θα δημιουργήσουμε και γραφειοκρατία τον εαυτό μας. Και Κάθε φορά που ένας Ελίας κάπου στην Ευρώπη κάνει κάτι λάθος ε, και πουλά ε, προϊόντα που θα είχε πάνω την ευρωπαϊκή ετικέτα, κάποιος ε, θα το μάθει αν γίνει κάτι λάθος και θα φταίει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, θα λένε, α δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτήν την οικολογική ετικέτα, ας μην το κάνουμε λοιπόν. Ε, και έχω πρόβλημα με τις ημερομηνίε. Εγώ προτιμώ τις ημερομηνίε εκφόρτωσης από τις αλλιεύσεις, αλλά γενικά είμαι υπέρ της διαφανές, αλλά δεν καταλαβαίνω πως οτιδήποτε από αυτά εγγυάται ότι πραγματικά εγγυόμαστε στον καταναλωτή Κοιτάξτε, μπορεί να παίρνουν το πιο φρέσκο ψάρι, αλλά είναι και το πιο υγιές το ψάρι. Δηλαδή, ε, μπορεί το σχάρι, να συγκρίνουμε ένα αποψυγμένο ψάρι με ένα ψάρι που ελεύθηκε πριν λίγες μέρες, αλλά σε ένα πολύ ζεστό κλίμα. Ε, δηλαδή, η προφανή σύγκριση είναι να έχουμε δεδομένα όπως έχουμε για κάθε ζώο που πάει στο σφαγείο. Αυτή είναι η προφανή σύγκριση. Νομίζω ότι δεν γίνεται. Μάλιστα. Σαν τη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τηλεγραφικά να πω ότι θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση, ότι πρέπει να θεσπίσει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των λειτουργιών ε, των οργανώσεων παραγωγών και της γεωργίας. Επίσης πρέπει οι οργανώσεις παραγωγών ε, να ε, τηρούν τις υποχρεώσεις της ποιότητας και πρέπει να δίνονται και πιο κατάλληλες πληροφορίες στον καταναλωτή αλλά και για να προωθηθεί η πώληση του νοπού ψαριού και σε ό,τι αφορά την επισήμανση νομίζω ότι είναι καλό, καλή οικολογική ετικέτα για συγκεκριμένα αλλιεύματα και θα μπορούσαμε επίσης να θέσουμε την δυνατότητα μιας ετικέτας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη Γεωργία και την Ελία που σέβεται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντεπίπερα από την Κομισιόν. Thank uh, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Στίβενσον ε, για την έκθεσή του. Επίσης είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι διαπιστώνω ότι υπάρχει συνολική υποστήριξη για το πακέτο των προτάσεών μας. Ε, σημειώσαμε τις ε, προτινόμενες τροπολογίες και δημονούμε να παραλάβουμε και άλλες Φυσικά για κάποια ζητήματα παρατηρώ διάσταση απόψεων, αλλά αυτό είναι προφανές. Επίσης υπάρχουν ε, κάποια άλλα σημεία για τα οποία ζητάτε μεγαλύτερη ενημέρωση για ιδιαίτερα τεχνικά ζητήματα. Ίσως δεν είναι το σωστό βήμα. Νομίζω διμερώς με τον κύριο Στίβενσον, με τους σκιώδεις εισηγητές θα μπορούσαμε να σας ενημερώσουμε. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ, κύριε Στίβενσον, να κλείσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα πολλά μέλη της Επιτροπής Αλίας που σχολίασαν. Με βοηθείτε πολύ με τα σχόλιά σας και επιθυμώ να ακούσω και τις λεπτομερείς απαντήσεις της Κομισιόν στις πολλές λεπτομερείς ερωτήσεις που της υποβληθήκαν για ορισμένα από τα ουσιαστικά θέματα που έθεσαν μέλη της Επιτροπής μας. Πρώτα για την ε, οικολογική επισήμανση. Γνωρίζω ότι συμφωνούμε, ε, διαφωνούμε επί της αρχής της Αβέλα. Ίσως μπορώ να καθισχάσω ορισμένους φόβους που εκφράστηκαν από τον Κρίς Τέιβης, διότι αυτό που προτείνω εγώ είναι για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα διαφορετικά 63 σήματα οικολογική συμμόρφωση, ξέρω εγώ, πέστε τα όπως θέλετε, τα eco σε αυτά, που όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφός μα ορισμένα δεν είναι παρά απάτη ορισμένων οργανισμών, για να, μπορούμε να, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλη αυτή τη σύγχυση που προκαλούν στους καταναλωτές, εγώ προτείνω ένα οικολογικό σήμα το οποίο θα ε, στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό να αναλυφθεί εργολαβικά, ας πούμε από το FMC, αυτό δηλαδή που υπάρχει ήδη, αλλά θα είναι μια υπηρεσία η οποία θα πληρώνεται. Δεν θα υπάρχει λοιπόν επιβάρηση του κοινοτικού προπολογισμού. Η ε, Κομισιόν θα προτείνει τα κριτήρια βασισμένα στα κριτήρια του ΦΑΟ και άλλα παρόμοια κριτήρια που ισχύουν για, άλλες, ε, για άλλα σήματα του αγροτικού τομέα. Επομένως, άλλοι οι οποίοι θέλουν να εξάγουν προϊόντα αλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, ε, αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σήμα, να σέβονται ακριβώς τα ίδια κριτήρια τα οποία θα ελέγχονται από το AMC και το SAC. Αυτό, αυτή είναι η ιδέα Έχω κάνει συζητήσεις με το MSC για το θέμα αυτό. Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο αναγνωρίζουν την αξία των ε, επισημάνσεων του MSC και εγώ δεν έχω αντίρρηση, τους είπα, να είναι το δικό τους λογότυπο δίπλα στην ευρωπαϊκή σημαία, ώστε να έχει απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα ο καταναλωτής ότι πρόκειται για βιώσιμο προϊόν το οποίο έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο οργανισμό. Δεν προτείνω δηλαδή καμία τεράστια γραφειοκρατία τώρα ε, που να προκύψει από, τις, την Επιτροπή, να, να δηλαδή στα γραφεία της Επιτροπής. Προτείνω να αναλυφθεί εργολαβικά από ανεξάρτητο οργανισμό, να γίνεται δηλαδή ο έλεγχος και η χορήγηση αυτού του σήματος. Ελπίζω με τον τρόπο αυτό να καθησυχάσω όπως είπα ορισμένους από τους συναδέλφους που εξέφασαν αμφιβολίες διότι έχει προκριθεί όντως κάποια σύγχυση. Για τις απορρίψεις τώρα. Η δική μου άποψη για τις απορρίψεις ελπίζω να μπορέσουμε να, τις, να, να αποφύγουμε τα παρελκόμενα αλλιεύματα με χρήση τεχνολογικών μέσων. Αλλά μοιραία κάποια είδη τελικώς θα λέγονται και θα εκφορτώνονται ακόμα και με την απαγόρευση των απορρίψεων. Και εφόσον πρόκειται για μη εμπορικά είδη ή για ηχθίδια που δεν θέλουμε να μπουν στην αγορά, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί αγορά, θα δίνεται στους κυβερνήτες των σκαφών ε, μια στοιχειώδης αποζημίωση, διότι ε, για να τους αποζημιωθούν για το καύσιμο που ε, κατανάλωσαν για να φτάσουν μέχρι την σειρά να τα εκφορτώσουν και τα, από τα, υπόλοιπα χρήματα να μπαίνουν σε ένα ταμείο το οποίο θα χρησιμοποιείται, τα χρήματα το οποίο θα χρησιμοποιούνται για ε, διατήρηση των ειδών. Εφόσον είναι εμπορεύσιμα τα ίδια αυτά, τότε που αλλιεύονται θα μπορούν να διοχετεύονται στην αγορά, σε τιμές αγοράς, αλλά από τα χρήματα αυτά που θα λαμβάνονται από την αγορά αυτή θα δίνεται μόνο ένα μέρος ως αποζημίωση στον κυβερνήτη και τα υπόλοιπα θα καταλήγουν σε ένα ταμείο διατήρησης και το υπόλοιπο θα ε, το αναλαμβάνει η οργάνωση παραγωγών αφού υπάρχει ενδεχόμενο ορισμένα πελαγικά είδη να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως δολώματα και επομένως πρέπει να ψυχθούν, πρέπει να μπουν σε ψυγεία δηλαδή. Άρα ορισμένα από τα χρήματα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίζουν το κόστος της αποθήκευσης. Εκεί που μιλούμε για τις ημερομηνίες αλίευσης και εκφόρτωσης μετά από πολλές συζητήσεις με τον αλλιευτικό κλάδο που μου είπαν γιατί τα έχω ξαναπεί εδώ στην Επιτροπή μας αυτά, ε, τους είπα, εάν επιμένετε υποχρεωτικά για την αλίευση, η τράτα που έχει βγει για ψάρεμα 5-6 μέρες και έχει βάλει το ψάρι σε πάγο, θα πρέπει να βγει στην εφόρτωση και να πει ότι είναι 5 ε, ημερών. Ενώ ένας που κάθεται την, ε, σε ένα μικρό σκαφάκι και ψαρεύει με το καλάμι ή την πετονιά ένα ψάρι θα μπορέσει να το βγάλει, παρόλο που το έχει αφήσει τον ίδιο όλη την ημέρα, να το βγάλει το βράδυ και να πει «Α, κοιτάξτε, είναι φρέσκο το ψάρι», ενώ το άλλο που είναι των 5 ή 6 ημερών θα είναι για τον καταναλωτή πλέον ε, όχι φρέσκο. Και μάλιστα και η ψαράδες του Πόρτο Νόβο στη Γαλλικία που είναι μικρή κλίμακα ψαράδε, μου είπαν ότι όντω συμφωνούν ότι υπάρχει εδώ κάποια ανισότητα. Όσο λοιπόν μπορούμε να βάλουμε την ημερομηνία τη αλήσευσης ω εθελοντική μου είπαν είναι πλεονέκτημα αυτό για μας. Αν μπορούμε να φέρουμε για την, μιλώ, για τη μικρή αλία το ψάρι να το βγάλουμε αμέσως την ίδια μέρα έχει καλώς. Αλλά να είναι εθελοντικό, ενώ υποχρεωτικό να, υποχρεωτική μάλλον να είναι η ημερομηνία εκφόρτωσης. Αυτός είναι ο λόγος που ε, έκανα την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι κάλυψα τα πιο πολλά ουσιαστικά θέματα. Αλλά ευχαρίστω να συναντηθώ ξανά με τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες να τις ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Λοιπόν, ε, νέα προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 12 Απριλίου το μεσημέρι. Και να περάσουμε στο τελευταίο σημείο που έχουμε για σήμερα το πρωί, γιατί έχουμε ακριβώ μισή ώρα. Αλία με τρεις και παραδοσιακή και τη μεταρρύθμιση και πολιτικής. 12 και 13. Τι είπα, λέει ο πρόεδρος. 12, 12. 12 Απριλίου το μεσημέρι. Αν είπα 13, συγγνώμη. Λοιπόν, σημείο 12. Στη, ε, τον Ιανουάριο είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και επίσης το Φεβρουάριο είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων. Δεν υπήρχε βέβαια χρόνος ε, για την ε, υλοποίηση την ολοκλήρωση της μελέτης με τον κύριο Φεραίρη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα να συμπληρώσουμε αυτή τη συνεδρία του Φεβρουαρίου και θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Φεραίρα έχει το λόγο και κατόπιν να μου πείτε ποιο θα πάρει το λόγο για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε και το χρόνο. Ευχαριστώ. Είδα εδώ ότι ήδη κάποιοι ζητούν το λόγο. Εγώ έκανα παρουσίαση του εγγράφου στην προηγούμενη ε, συνεδρίαση και ήδη στι προηγούμενε δύο συνεδριάσει είχα προσεγγίσει κάποιε από τι πτυχέ κλειδιά ε, του εγγράφου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χάσουμε περισσότερο χρόνο και ε, βάλαμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη γιατί οι συνάδελφοι που δεν μπόρεσαν να τοποθετηθούν να μπορέσουν τώρα να πάρουν το λόγο. Έτσι λοιπόν εγώ δεν θα πω άλλο. Μάλιστα ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο κυρία Φράγα. εγώ θα επεκταθώ πάρα πολύ γιατί μίλησα τις προάλλες για το θέμα, απλώς ε, εκμεταλλευόμενη και όσα είπε η κυρία Ρόντουστ προηγουμένως ε, και όσα λέει ο κύριος Φεραίρα στην έκθεση, να συζητήσουμε και πάλι το θέμα του ορισμού της ε, ε ε, της ή όπω θέλετε να την αποκαλέσουμε. Το σκεφτόμουν το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα ήταν ε, καλό να συμφωνήσουμε. Ήδη έκανα και μια σχετική πρόταση σε δύο παραμέτρους που θα μπορούσαν να είναι εναλλακτικέ. Και εγώ νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο θα κάλυπταν αρκετά καλά μια αριστεχνική αλία, τι μπορεί να είναι. Και όπως πάντα θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη το μήκος ε, του σκάφους, 12 μέτρα ή θα το δούμε. Για να μην ανοίξουμε περαιτέρω τη συζήτηση, θα μπορούσαμε να το αφήσουμε στα 12 μέτρα μήκος, αλλά υπάρχει και άλλη μία παράμετρος ε, που ε, μα δείχνει πάρα πολύ καλά τι είναι η μικρή ελία. Ε, και ε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε πόσο παραδείγματος χάρη ε, διαρκεί ΕΕ, η παλήρια. Νομίζω ότι αν μιλάμε για 24 ώρες αυτό θα είναι κάτι ενδεικτικό. Γιατί αν συζητήσουμε με τον κλάδο και με την Κομισιόν τον ορισμό που υπάρχει στο δασικό κανονισμό για την αριστεχνική αλία, κάποιος κατανοεί απόλυτα ότι μπορεί να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ στόλου που πραγματικά είναι αριστοτεχνικό λόγω της διάρκειας ε, των παλιωρών να μπορεί να έχει στα σκάφη ένα ε, μέτρο ε, περισσότερο ή λιγότερο μήκο. αλλά αυτό είναι αντισκαφών που ε, παραδείγματος χάρη αλλιεύουν ε, το ίδιο είδος και νομίζω ότι η παράμετρος της διάρκειας της παλήρες 24 ώρων μπορεί να είναι ε, κάτι ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να είναι εναλλακτικό κριτήριο του μήκους των 12 μέτρων. Εγώ ανέφερα αυτή την ιδέα και σε οποιαδήποτε περίπτωση νομίζω ότι μπορούμε να τη συζητήσουμε και Ούτε πιστεύω ότι είναι καλό να φτάσουμε σε ένα πολύπλοκο ορισμό εγώ προσπάθησα να βρω δύο αντιπροσωπευτικά κριτήρια, ένα που ήδη έχουμε και αυτό που σας είπα σε σχέση με τις 24 ώρες ε, για τη διάρκεια της βαλήριας, για να ε, μπορέσουμε να προσδιορίσουμε καλύτερα τι είναι αυτή η μικρή παράκτια αλία. Δεν θέλω τώρα να μπω εγώ σε άλλο θέμα, ε, στην εκθέση του κυρίου Φερέιρα αλλά ήθελα να καταθέσω αυτή την άποψη εδώ δημοσίως και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έγγραφο εργασίας επικρίνει σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και νομίζω ότι είναι άδικο αυτό. Δεν έχω και πάρα πολύ καιρό εδώ στην Επιτροπή Αλία, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω η θέση των αλλιών τη Αλία σε μικρή κλίμακα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τι εθνικέ αποφάσει, αποφάσει των κυβερνήσεών του. Αν επιθυμούν να βοηθήσουν λοιπόν του μικρού αλίες, οι κυβερνήσεις, κυρίω ε, στι περιοχέ όπου έχουμε ποσοστό και τάξη, α του δώσουν μεγαλύτερο μερίδιο. Θέλω να ακούσω και την άποψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ε, κα, κατακρίνεται Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ πρωτίστω πρέπει να είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ε, όλη αυτή η ιδέα των μεταβιβάσιμων ε, παραχωρήσεων ε, σίγουρα δέχεται πολύ ισχυρέ επικρίσει, αλλά βλέπω μέσα στο έγγραφο εργασία πω ουσιαστικά προτείνεται η πρόσβαση στου πόρου να υπάγεται σε ένα ενιαίο σύστημα. Ε, τα TFC όμω ε, δεν είναι ένα ενιαίο σύστομο, δηλαδή μπορεί να σχεδιάσει κανείς μεταβάσιμες παραχωρήσει σε επίπεδο κρατών μελών, τόσο να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικέ προτεραιότητε και η κατάσταση επιτόπου. Αν θέλετε να προστατεύσετε την αλία μικρή κλίμακα, μπορείτε να σχεδιάσετε ε, με τα TFC ή να εφεύρετε ένα οποιοδήποτε σύστημα. Υπάρχουν διάφορα, διάφορες μορφές, αν θέλετε, μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, και διακρίνω ένα φόβο, ίσω και δικαιολογημένο, δεν τα καταφέρουν τα κράτη-μέλη και ότι θα είναι ολέθριο ο σχεδιασμό των TFCs ε, και έχουμε τέτοια κακά παραδείγματα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ενιαίο το σύστημα, είναι ευέλικτο συγγνώμη, και τα κράτη-μέλη σχεδιάζουν βάσει των προτεραιοτήτων του ε, τα TFCs. Για την περιφερειοποίηση, πάλι στο κανονισμό για την κοινή αλληλευτική πολιτική δεν υπάρχουν πολλές διατάξεις που να περιγράφουν την μορφή που θα πάρει αυτή η περιφερειοποίηση Όπω ακούσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως ε, ε, ανέκαθεν ήταν ανοιχτή. Δηλαδή, εγώ πάντοτε έβλεπα ότι ξεκινούσα από τη βάση, ξεκινούσαμε από τη βάση και αποφασίζαμε. Μπορούμε να θεσπίζουμε κριτήρια και να πούμε να οι περιφερειακοί οργανισμοί τώρα θα αποφασίσουν. Γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ σε ένα περιοχή. Κάποιοι οργανισμοί λειτουργούν πολύ καλά, είναι καλά οργανωμένοι και είναι έτοιμοι να αναλάβουν ε, διευρυμένε αρμοδιότητε. Τα λέγατε κι εσεί για τη Σκοτία κτλ είναι ένα παράδειγμα όπου ο ντόπιο οργανισμό μπορεί να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκινάμε από τη βάση. Και θέλω να μου πει ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι που λείπει από τον κανονισμό, να μου πει λοιπόν με ποιο τρόπο θα αντιδράσει σε, ως προς αυτό το θέμα, δηλαδή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους οργανισμούς ε, που είναι έτοιμοι για ε, μεγαλύτερη χώριση αρμοδιοτήτων και τους υπολείπους. Δηλαδή θα είναι θετικές οι αντιδράσεις πάντοτε ε, ή θα αντιδράσουν και θα προσπαθήσουν παρόλα αυτά, παρά τα όσα υπόσχονται να έχουν κεντρικό έλεγχο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεβίτ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ρουσέτ. Μπέσετ, συγγνώμη, ε, πιστεύω ότι το έγγραφο εργασίας ε, του κυρίου Φερέιρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, διότι μας προσφέρει δύο εναλλακτικές οδούς για να σημειώσουμε πρόοδο στο συνολικό προβληματισμό μας για την μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Δύο εναλλακτικές οδούς λοιπόν. Πρώτον, ως προς τον ορισμό της μικρής αλληλεία, παράκτες αλληλεία, αεριστεχνικές αλληλεία, όπως και αν την χαρακτηρίσουμε γιατί υπάρχουν πολλοί επιθετικοί προσδιορισμοί Πάντω, ε, ποιο είναι ο κοινό προνομαστή. Ε, μέσα στο έγγραφο εργασία του κ. Φερέιρα απαριθμούνται διάφορα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό και η δεύτερη λύση που μα προτείνει ο κ. Φερέιρα είναι τρόπου ε, με του οποίου θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε την μικρή αλία η οποία είναι απαραίτητη κατά γενική αποδοχή όχι μόνο για τη διατήρηση των θέσεων εργασία αλλά και για την προστασία των αλληλευτικών πόρων. Ε, ως προς τον ορισμό, ε, ε, πρόκειται για μια ουσιαστικότερη δυσκολία. Ε, περί τίνο πρόκειται. Ε, Κυρίως πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιον θα εφαρμοστούν τα ειδικά μέτρα, αν τελικά θεσπιστούν ειδικά μέτρα για αυτού του είδους ε, την αλία. Η πραγματικότητα ε, στον κλάδο αυτό ε, είναι, διαφέρει φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα. Αν έχω σωστά στοιχεία, η αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των δύο εγκεκριμένων κριτηρίων, δηλαδή το μήκος του σκάφους άνω ή κάτω των 12 μέτρων και η προσφυγή ε, σε με ε, αλλιευτικό ε, εξοπλισμό ειδικό για τη μικρή αλία. Δίνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10% ποσοστό της μικρής αλίας στο σύνολο του κλάδου και κυμαίνονται τα ποστα 10, 11, 12% και σε ορισμένες περιοχές μιλάμε για το 75-80% των αλλιευτικών σκαφών. Η κυρία Δαμανάκη μας είπε ε, ότι ε, το θέμα της εραστεχνικής αλλίας αγγίζει το 80% του στόλου. Λοιπόν, τι ισχύει από όλα αυτά, ποια είναι τα σωστά αριθμητικά στοιχεία, γιατί πράγμα μιλάμε. Είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτή η έκθεση του κυρίου Φερέρα ούτως ώστε να υιοθετήσουμε μια ορθότερη προσέγγιση, είναι και να ξέρουμε πώς, ποιο προσανατολισμό θα ακολουθήσουμε κατά την εκπόνηση των πολιτικών μας. Απαριθμη, ε, ε κριτήρια και οι παράμετροι σίγουρα θα είναι ένα συνοδήλευμα όλων αυτών των στη γέννη. Η κυρία Φράγκα μα μίλησε και για την ε, διάρκεια τη αλληλευτική προσπάθεια πέρα από το μέγεθο ε, των σκαφών, το μήκο και την ισχύ του κινητήρα. Ε, υπάρχει αυτό. Επίση υπάρχουν τα ίδια αλλία με διαφορετικέ ε, περιβαλλοντικέ επιπτώσει, επιπτώσει επί των φυσικών πόρων και διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό ρόλο κτλ. Τα, τα διάφορα ίδια αλλία λοιπόν. Τέλο πάντων, για να μην πολυλογώ, ε, πώ θα οριοθετήσουμε την ε, αλία μικρή κλίμακας. Θα προκαλέσω λίγο, αρχίζοντας ε, την συζήτηση, ε, θα πω ότι η μικρή αλία δεν είναι αυτή που γίνεται με το δίχτυ. Νομίζω ότι είναι καλό εφαλτήριο η έκθεση του κ. Φεραίρα για να προβληματιστούμε για τον ορισμό. Δεύτερον, προτείνει διαφοροποιημένη προσέγγιση ο κ. Φεραίρα, ειδικό καθεστώ συγκεκριμένα για τη μικρή αλία, δηλαδή ένα είδο θετική διακριτική μεταχείριση υπέρ αυτού του υποκλάδου. Ε, τώρα, δεν θα θέλαμε... Ε, ε, να αποσυνδέσουμε τι πιθανέ ε, αποκλείς εξαιρέσει για την ε, αλία μικρή κλίμακος, να τι αποσυνδέσουμε από τι αρχέ της μεταρρύθμισης τη κοινή αλλιευτική πολιτική, διότι αυτέ οι αρχέ κατά τη γνώμη μα είναι ο βέλτιστος τρόπο για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα του κλάδου αυτού. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να προστατεύσουμε την αλία μικρή κλίμακος. Έτσι θα έχουμε τι καλύτερε πιθανότητε σε αυτόν τον αγώνα για να προστατεύσουμε προστατεύσουμε την αλία. Ε, μιλάμε για την αιρεσιμότητα της βιώσιμης αλίας με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, με την, ε, το στόχο ε, των μηδονικών απορρίψεων, με τις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις και παραχωρήσεις που θα είναι το τέλος της μικρής αλίας, η συνδιαχείριση από όλου του εμπλεκόμενου φορεί, όλα αυτά τα κριτήρια είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα τη αλληλεία μικρή κλίμακα. Ε, τη σήμερον ημέρα, το τονίζω, ε, θα πρέπει να διεκδικηθούν σε αυτόν τον αγώνα και οι κανόνε ε, του παιχνιδιού θα είναι ακριβώ αυτά τα κριτήρια που ισχύουν γενικότερα για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Ευχαριστώ, κύριο Καντέκ. Έλειπα, λέει ο κ. Κατέκτη, την προηγούμενη φορά που το συζήτησα το θέμα και μπορούσα να συμμετάσχω και τώρα που ε, συζητείται η έκθεση Φεραίδα τον οποίο συγχαίρω για την ποιότητα της εργασία του, παρόλα αυτά φοβούμε και το έχω πει εδώ και χρόνια, από την αρχή δηλαδή της παρούσας θητείας, ότι το να καταλήξουμε σε ορισμό στο πανευρωπαϊκό επίπεδο για την βιοτεχνική αλία, η μικρή κλίμακα αλία, μου φαίνεται αδύνατον. Δεν είναι η ίδια ε, η αλία αυτή στις ακτές της Μάχης ή στη Μεσόγειο ή στην Βαλτική. Και εν προκειμένου ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μένα είναι, τι να πω, τι θα πει 12 μέτρα στην Βρετάνη ψαρεύουν ένα κοχύλι του Αγίου Ιακώβου με υποδειγματικό τρόπο εδώ και δεκαετίες είναι βιώσιμη αλλή αυτή παίρνουν ε, ε, ε, σκάφη της τάξης των 8,5 μέτρων και με παρασυρώμενα εργαλεία. Επομένως ο ορισμός για μένα είναι απολύτως απαράδεκτος. Ο Ζαό Φερέιρα προσπάθησε να καταλήξει σε κριτήρια που να μπορούν να καθορίσουν τη μικρή κλίμακα αλληλεία είναι το μέγεθος, είναι τα αλληλευτικά εργαλεία, το είπε αυτό η κυρία Φράγα. Επαναλαμβάνω ότι η μικρή κλίμακα δεν είναι η ίδια σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα κοινό ορισμό. Εγώ νομίζω μάλιστα ότι αυτό είναι αδύνατο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η βιοτεχνική αλία, το είπε και ο κ. Μπεσέ προηγουμένω, είναι ό,τι δεν είναι βιομηχανική αλία. αφού δεν θα μπορέσουμε. Καλύτερα να ορίσουμε κάτι άλλο. Στην Ελλάδα μπορεί η, η, η ε, ε, μικρή κλίμακα μπορεί να είναι με, ένα, με μια βάρκα 4,5 μέτρα με δύο κουπιά. Ε, παρβάρω λίγο, αλλά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Στη βρετανη είπα είναι 8,5, 10, 12 μέτρα. Είναι λοιπόν πολύ διαφορετικά. Θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε έναν ορισμό της μικρής κλίμακας ή παραδοσιακής αλίας. δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα αυτό το κριτήριο της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 12 μέτρων. Δεν μπορώ να το δεχτώ λοιπόν. Δεν έχω βέβαια και καμιά άλλη απάντηση για να σας πω η βιοτεχνική αλληλεία είναι αυτό. Θα προτιμούσα να πούμε τι δεν είναι. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Άλλωστε, στην έκθεση του Ζωάου Φερέιρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μηχανισμός αντιμετώπισης επίγουσων καταστάσεων, η στήριξη της μικρής κλίμακας αλίας κλπ. Ευχαριστώ κύριε Καρέκ. Μιλάνα. Η κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ. Η έκθεση του συνάδελφου Ζωά παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, πολύ σημαντικές ε, γιατί έχουμε και τον ορισμό ε, της ε, αεροστεχνικής αλίας, ε, γιατί είναι πολύ περιοριστικός ο ορισμός που, περιορι... που παρουσιάζει η, Επιτροπή. Ε, το ένα θέμα οδηγεί στο άλλο. Η οικολογική, επιστημονική, η οικονομική βιωσιμότητα και η τοπική βιωσιμότητα είναι όλα ενωμένα. Οι βασικές αρχές ε, της μεταρρύθμισης αποτελούν τη βάση. Αλλά κατόπιν, αν δεν αναγνωριστούν ε, όλα τα θέματα, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, αν δεν υπάρχει προστασία, αν δεν υπάρχει ειδική μεταχείριση, δεν θα μπορέσουμε ε, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει η αεραστεχνική γεωργία ή η καλή εκτροφή μαλακίων ή ε, εκτατική καλλιέργεια. Αυτά θέλω προσθέσω από τη σκοπιά της Επιτροπής Ρέτζη και επίσης ε, το να λέμε ότι η αεραστεχνική ελία είναι μια οικογενειακή ελία πρέπει να το λάβουμε υπόψη, πρέπει να υπάρχει και αναλλαγή των γενεών και αυτό είναι ένας τρόπος ε, να υποστηρίξουμε αυτή την εναλλαγή των γενεών, ε, γιατί πολλές φορές ε, στην αριστεχνική αλία ένα σκάφος είναι ένα άτομο και ένα άτομο είναι μια οικογένεια και έχουμε οικογένειες που εξαρτώνται πάρα πολύ από την αλία και αυτό συμβαίνει στη δική μου χώρα. Ευχαριστώ, η κυρία Λουβέν. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να προσθέσω μόνο ένα στοιχείο και πιστεύω ότι ο κύριος Ντέιβις ε, το ανέφερε εν μέρη. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό αυτά που προτείνεται κύριε Φερέιρα ε, είναι ούτως ή άλλως ήδη θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Ζητάτε μέτρα στήριξης για κατεπήγοντα περιστατικά, όταν ε, ε, προβλέπετε περιόδους ε, ανάπαυσης, υποστήριξη προς τους αλληλείς. Στη Σουηδία ήδη συμβαίνουν αυτά. Ε, ε, τώρα σε σχέση με την πρόσβαση σε αυτή την αλληλευτική ζώνη των 12 ε, μιλίων και η προτιμησιακή πρόσβαση για τους μικρούς αλληλείς, και αυτό συμβαίνει, δηλαδή μπορεί η κυβέρνηση δικαιούται να επιφυλάξει διαφορετική μεταχείριση για τα διάφορα υποτμήματα του κλάδου. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη μικρή αλληλεία, συγγνώμη, ανάμεσα στις βόρειες και στις νότιες χώρες και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς την περιοχή ζώνη των 12 μιλίων για να ορίσουμε την ε, αλληλεία μικρή κλίμακος, τουλάχιστον όχι στη Σουηδία, ίσως ε, στη Νότια Ευρώπη. Πάντω η κυβέρνηση έχει αυτό το δικαίωμα και επιφυλάσσει διαφορετική μεταχείριση ε, για τα διάφορα υποτμήματα του κλάδου. Ο κ. Πάντο Κούπερ τώρα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την πρωτοβουλία του. Όπως σας είπα και την περασμένη φορά είναι πολύ σημαντική η έκθεση γιατί η αλία μικρής ε, ε, κλίμακας ε, εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ αρχής θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί αναφέρθηκαν κάποιοι σε διάφορα ποσοστά. Ε, υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Όποιον ορισμό και αν χρησιμοποιήσει κανείς, ας πάρουμε το δικό μας, έχουμε διαφόρων διάφορα επίπεδα ε, αλληλείας μικρής ε, κλίμακας ε, ανακράτος μέλος, δηλαδή κάτω, παραδείγματος χάρη των 100 σκαφών, Α, συγγνώμη, τα ποσοστά δηλαδή των μικρών σκαφών ε, στον συνολικό στόλο διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Μιλήσατε για 80%, μπορεί να είναι και 99% και 100%. 80% ε, των σκαφών βάσει του δικού μας ορισμού ε, υπάγονται στην κατηγορία μικρής αλίας και άρα νομίζω ότι όλες μας οι πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν και να καλύπτουν επαρκώς την βιομηχανία την αλία μικρής ε, κλίμακος. Ε, αυτά εν γέννη και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία από τον ιολόγιό μας να σας τα προμηθεύσουμε ευχαρίστως. Ένα μεγάλο τμήμα του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάγεται στον ορισμό της αλίας μικρής κλίμακος όπως τον προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το θέμα του ορισμού που σας έλεγα και τις προάλλε, είναι πάρα πολύ σημαντική και περίπλοκη αυτή η συζήτηση. Η Επιτροπή από πλευρά τη έχει κάνει πολλές τέτοιες συζητήσεις συζητήσει τα προηγούμενα χρόνια για να προετοιμάσουμε παραδείγματο χάρη χρηματοοικονομικά μέσα που πλέον χρησιμοποιούνται, ε, συζητήσει εν ώψη τη μεταρρύθμιση και αποφασίστηκε μετά από όλε αυτέ τι συζητήσει να διατηρήσουμε αυτόν τον ορισμό για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί πάντοτε Υπάρχει ένα παζάρι ε, και όλοι προσπαθούν να συμπεριλαμβάνουν όλα ε, και πιο τεχνικές διατάξεις στον γενικό κανονισμό και προσπαθούν να προλάβουν τις ιδιαιτερότητες του ε, στόλου τους. Ε, ο συνδυασμός ε, του κριτηρίου του μεγέθους και το είδος του εξοπλισμού σταθερού ή παρασυρώμενου νομίζω πρέπει να συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε ορισμό και στην καθημερινή πρακτική όπως βλέπουμε και στο Ταμείο Θάλασσας και Αλίας και νομίζω θα συμφωνήσουν τα περισσότερα κράτη-μέλη και με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε μεγαλύτερα ε, προβλήματα. Ε, on 24 hour. Ε, όταν ε, Όποιο ε, καινούριο στοιχείο εισαγάγουμε στον ορισμό συνεπάγεται περισσότερα μέτρα ελέγχου και εποπτείας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ε, θα ήθελα να διευρύνουμε και τη συζήτηση για τον ορισμό για να κατανοήσουμε από πλευράς πολιτικής τι είναι εφικτό. Είπαμε τα κρατη λίγη και είπατε και σωστά, ότι έχουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών ε, στα πλαίσια της χάραξης της εθνικής τους πολιτικής. Θα ήθελα να σε εξηγήσω πώς λειτουργεί το σύστημα της κατανομής των ποσοστώσεων. Κατόπιν πρότασή μα, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο ε, προσδιορίζει τα τάξη και τις αλληλευτικές ε, προσπάθειες. Ε, στη συνέχεια, αναπόθεμα υποδιαιρείται το σύνολο βάσει της κλίδας κατανομής της περίφημης και στη συνέχεια είναι μάλλον εθνικό θέμα. Δηλαδή, το κράτος μέλος αποφασίζει ποιος θα πάρει τι από αυτή την συνολική ποσόστοση και ακόμη και σε εκείνο το γύρο, δηλαδή στην κατανομή των αλληλευτικών δυνατοτήτων, κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιεί δικό του ορισμό. Η Ισπανία έχει δικό της ορισμό ε, υπέρ ή κατά παραδείγματο χάρη ε, συγκεκριμένων ειδών αλληλείας, ε, δηλαδή τα ίδια τα κράτη-μέλη δημιουργούν αυτό το περιθώριο ελιγμών και έχουν διαφορετική μεταχείριση για διάφορα τμήματα του στόλου τους. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει για να να αυτά τα στοιχεία που θα συνυπολογίζονται κατά την κατανομή. Αλλά εν τέλει είναι εθνικό το θέμα, θέμα εθνική αρμοδιότητα και είναι καλό που έχει το περιθώριο κάθε κράτο μέλο. Ε, είναι σωστό που η Φινλανδία δεν χρειάζεται να ακολουθεί την ίδια λογική όπω το Βέλγιο κατά τη χάραξη τη πολιτική τη. Ο ορισμό ε, πάντω έχει ε, περιορισμού ω προ την αξία του και γενικότερα έχει πολλού περιορισμού λόγω αυτών που σα είπα. Ο κύριο Ντέιβι μα μίλησε για τα TFC, τι παραχωρήσει δηλαδή ε, που ε, κατακρίνονται στην έκθεση μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό το σύστημα όπως το προτείνουμε αφήνει μεγάλο περιθώριο πάλι ε, ελιγμών για τα κράτη-μέλη για να κρίνουν βάσει των ε, δικών τους ε, αναγκών, των ιδιαιτεριοτήτων, την κατάσταση της αλληλεία στη χώρα τους, κατά πόσο χρειάζονται ρήτρες ή δικλείδες ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ θετικό που έχουν αυτό το περιθώριο τα κράτη-μέλη. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με κάτι για το οποίο επιμείνατε κι εσείς και το έχουμε ξανασυζητήσει προηγούμενες συνεδριάσεις. Είπαμε ότι λέει για την πολιτική διατήρηση, συντήρηση του αποθέματος, ε, ε, δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε η μικρή αλία να είναι πιο βιώσιμη ή πιο φιλική περιβαλλοντικά. Ε, δεν θέλουμε για την πολιτική διατήρηση των αποθεμάτων να ισχύουν δύο μέτρα και δύο στάθμα κοινά. Θα πρέπει να είναι για όλους και μην ξεχνάτε ότι αλλιεύουν παράκτη κοντά στις ακτές αυτά τα σκάφη. Οπότε για το θέμα της προστασίας των πόνων τη αναπαραγωγή. Ε, και τα λοιπά θα πρέπει να είναι ίσως και πιο αυστηρά τα κριτήρια. Σε κάθε μία περίπτωση όμως δεν προτείνουμε διαφοροποιημένο καθεστώς. Τελευταία παρατήρηση, παρότι δεν αναγνωρίζεται αυτό ε, σε όλα τα, ε, στην έκθεση, έχουμε και τον βασικό κανονισμό όπου προβλέπονται τα περιτύευσης. Έχουμε τον κανονισμό για το Ταμείο Αλίας και στους δύο έχουμε συμπεριλάβει ειδικέ διατάξει ε, με στόχο να υποστηρίξουμε την ε, αλία μικρή ε, κλίμακα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι για τα κριτήρια για την κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων σε μεταγενέστερο στάδιο θα δείτε ότι συμπεριλαμβάνουν ακριβώ την αλία μικρή κλίμακας και το άλλο είναι ότι ε, θα θέλαμε να είναι πιο εντατική η βοήθεια που προσφέρεται ε, εφ' εξής, ε, στην αλία μικρής κλίμακας. και ούτω ή άλλω οι επιδοτήσει θα είναι υψηλότερε από αυτέ που προορίζονται για την βιομηχανική αλία. Έχουμε πολλά επιμέρου στοιχεία μέσα στι προτάσει μα που δείχνουν ότι λαμβάνουμε υπόψη ιδιαιτερότητε αυτού του κλάδου. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φερέιρα για δύο-τρία λεπτά για να ολοκληρώσει και ευχαριστώ τους διερμηνείς που θα μας δώσουν πέντε λεπτά ακόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια και εγώ θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια σχετικά με όσοι υπόθηκαν. Καταρχήν το θέμα του ορισμού. Εγώ καταγράφω τη συνεισφορά που βλέπω εδώ για να αναζητήσουμε εναλλακτικού ορισμού στον ορισμό που προτείνει η Κομισιόν, αναγνωρίζοντα ε, βέβαια του περιορισμού αυτή τη τελευταία. Θεωρώ ότι είναι θετικό και νομίζω ότι είναι καλή συνεισφορά για αυτή τη συζήτηση που φυσικά θα πρέπει να συνεχιστεί. Η Κομισιόν μας λέει και έχει επιμείνει σε αυτήν την ιδέα εδώ και καιρό ότι τα κριτήρια που προτείνουν καλύπτει το 80% των σκαφών. Ε, περίεργος όμως δεν μας λέει ποτέ ποιος είναι ο όγκος των ηχθείων και ο, ο όγκος των συναλλαγών που εμπίπτει σε αυτό. Εγώ και ένα σύνολο συναδέλφων είχαμε ε, την ευκαιρία να στείλουμε μια γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό το 80% ε, των σκαφών ε, και αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι είναι σωστό το νούμερο της Κομισιόν δεν αλλιεύουν το 80% των πόρων. Στην αλήθεια αλλιεύουν ένα πολύ κατώτερο ποσοστό Δηλαδή ο όγκος των ψαριών είναι πολύ χαμηλότερος από το 80%. Τι σημαίνει αυτό, εγώ δεν ξέρω αν η Κομισιόν θα ξέρει αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω για το σύνολο ε, της Ευρωπαϊκής και για ορισμένα κράτη και για τη δική μου χώρα ότι το 80% των σκαφών αλλιεύουν έναν όγκο του συνολικού εκφορτώμενου ποσοστού ψεριών που μπορεί να φτάνει στο 100% είναι αυτό που γνωρίζω. Εγώ δεν ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη, όμως εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό ουσιαστικό αυτού του τμήματος του στόλου. Και πάντοτε η Κομισιόν το τονίζει αυτό, όμως ε, ο στόλος αυτός αλλιεύει ε, τη μειοψηφία των ε, ψαριών, δηλαδή Έχουμε ένα άλλο τμήμα του στόλου που είναι πιο λιγάριθμο αλλά αλλιεύει το μεγαλύτερο μέλος των πόρων. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο τμήματων του στόλου και να τη διαχειριστούμε διαφορετικά. Τώρα, σε σχέση με την ευελιξία του συστήματος των μεταβάσιμων λευτικών παραχωρήσεων που ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι. Δεν αξίζει εδώ ε, να εφευρίσκουμε ε, επιχειρήματα. Το σύστημα μπορεί να είναι ευέλικτο, συνεχίζει να είναι σύστημα και το θέμα δεν είναι εδώ να πούμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά το σύστημα αυτό και να υπονοούμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Το θέμα είναι αν επιτρέπεται ή όχι σε ένα κράτο-μέλο ότι για να πετύχει ορισμένου στόχου να χρησιμοποιήσει άλλε λύσει πέραν του συστήματο αυτού του TFC. Η πρόταση τη Κομισιόν δεν το επιτρέπει. Εμεί κατανοούμε ότι αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται, δηλαδή να χρησιμοποιούνται άλλα συστήματα. Και δεν υπάρχει νόημα εδώ να μιλάμε για ευελιξία. Από αυτή τη σκοπιά ευελιξία στην πρόταση τη Κομισιόν είναι μηδενική. Δεν υπάρχει καμία ευελιξία γιατί υποχρεωτικά υποχρεωτικά επιβάλλει ένα σύστημα το οποίο μάλιστα θα συμπεριλαμβάνει πολλά από αυτά που εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνονται μέσα στην έννοια της αλληλίας μικρής κλίμακας. Το θέμα που επίσης αναφέρθηκε σχετικά με το ρόλο των κρατών μελών. Και ο συνάδελφος Ντέιβις ε, και η συνάδελφος ε, Λοβίν το ανέφεραν. Ε, πράγματι, το κράτος μέλος έχει ρόλο να διαδραματίσει την υπεράσπιση τη Αλία Μικρή κλίμακα και μάλιστα σε αυτό συνεισφέρει και η αποκλειστική περιοχή των 12 μιλίων και γίνεται μια θετική αξιολόγηση αυτή τη περιοχή των 12 μιλίων και προτείνεται να σταματήσει να είναι παρέκκληση για να έχει μόνιμο χαρακτήρα και προτείνεται επίση διεύρυνση αυτή τη ε, περιοχή. δηλαδή υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, επομένως αφού υπάρχουν ε, θετικά αποτελέσματα αποτελέσματα, γιατί να μην παγιώσουμε αυτή την εμπειρία, γιατί να μην δώσουμε στα κράτη-μέλη περισσότερα από τα μέσα από αυτά που έχουν σήμερα για να υπερασπιστούν τη μικρή αλληλεία. Μηχανισμοί εκτακτή ανάγκη, ε, μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά αυτό που κατανοούμε ε, και τελειώνω, Πρόεδρε, είναι ότι δεν αρκούν. Δεν ε, μπορούμε, και αυτό είναι μια εκτίμηση γενική, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι έχουμε μια πολιτική η οποία είναι κοινή για ορισμένα πράγματα και δεν είναι κοινή για άλλα. Δηλαδή δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι έχουμε μια πολιτική η οποία καθορίζεται κεντρικά και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να σέβονται τους προσανατολισμούς πολιτικής αυτής, αλλά στη συνέχεια όταν μιλάμε για ορισμένο από το κόστος αυτής της πολιτικής, αυτό να το σηκώνουν τα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει με τους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης. Και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε εδώ να προβλέπονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, για να υποστηρίζετε αυτό το τμήμα του στόλου και να μην αφήνεται στα κράτη-μέλη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και ολοκληρώνω με το σημαντικό ρόλο που τα κράτη-μέλη έχουν εδώ εδώ και σε πολλούς άλλους τομείς. Αλλά ακριβώς γι' αυτό αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να προσανατολιστεί όχι ε, σε ένα όραμα συγκεντρωτικό, αλλά σε ένα όραμα αποκεντρωτικό και ε, δυστυχώς οι προτάσεις της Κομισιόν δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα, σας ευχαριστώ όλους, ο ευχαριστώ και τους Γερμανείς και στις 3 θα συνεχίσουμε με την ακρόαση για την περιφερειοποίηση στα πλαίσια της μεταρρύθμισης.